possiamo prendere posto. Μπορείτε να καθίστε. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας. Μετά θα ψηφίσουμε. Έχουμε μία ώρα για το σημείο 14 στην ημερήσια διάταξη που είναι οι ενεργειακές διευρωπαϊκές υποδομές και η συγητής είναι ο Κορέια Ντεκάμπος. Καλό σας απόγευμα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Σκιώδη εισηγητή για τη συνεργασία που μου προσέφερε. Να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο που ανέπτυξε και για την συνεργασία που είχαμε. Να ευχαριστήσω επίσης και το Συμβούλιο που είχε την δυνατότητα που μας προσέφερε να συμμετάσχουμε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών για θέματα ενέργειας το την προηγούμενη εβδομάδα στην, στην ε, Κοπενχάγη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια αντίδραση είναι απόλυτα αναγκαία για τα ενεργειακά θέματα. Η ενεργειακή πολιτική υποχρεώνει σε ένα πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς από αυτό που υπάρχει σήμερα για τους τρεις στόχους, κύριου τρεις στόχους της δικής μας ενεργειακής πολιτικής. Ασφάλεια ανεφοδιασμού, πρώτος στόχος. Δεύτερον, να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα και με προσιτές τιμές ε, του κόστους ενεργειακών προϊόντων και να υπάρξει και η εφορία, ενεργειακή εφορία προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο είναι το γενικό πλαίσιο. Η δική μας γνωμοδότηση στοχεύει στο να συμφωνήσουμε και να υποστηρίξουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια πρόταση που θεωρούμε ότι είναι λογική με κοινό νου για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας την άρση, την αντιμετώπιση των προσκομμάτων και εμποδίων, μεγαλύτερη συνεργασία των κρατών μελών, μεγαλύτερο άνοιγμα, προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, αύξηση της απασχόλησης και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με την πρώτη ανάγνωση. Η συμφωνία από στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο είναι κάτι που επιθυμούμε και θέλουμε να υπάρξει η αντανάκλαση στην τελική πρόταση της θέσης αυτής. Αυτή είναι τώρα η θέση και τι γίνεται με τις τροπολογίες, με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Θέλουμε να ενισχυθεί η συνιστόσα η ευρωπαϊκή, να έχουμε πιο αποτελεσματικά μέσα για, την υποδο... για τις υποδομές, για την προαγωγή μιας μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ εκείνων που εκμεταλλεύονται τα δίκτυα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και φυσικά αυτονόητο είναι ότι στην επιλογή των προγραμμάτων κοινού συμφέροντος η συνεργασία να διευρυνθεί ώστε να υπάρξει η συμπερίληψη και των εταίρων στα δίκτυα κατανομής ώστε να υπάρξει μια αλληλοσύνδεση δικτύων και αλληλουχία δικτύων. Οι εξουσίες απόφασης των περιφερειακών σωμάτων είναι θέμα της Επιτροπής και του Συμβουλίου προτείνουμε ενίσχυση του ρόλου της ΑΣΕΡ, της, ε, του συνδέσμου ρυθμιστικών αρχών της Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών, ώστε να υπάρξει η προώθηση αυτού του προγράμματος και η επιλογή προγραμμάτων, ώστε να έχουμε αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, ώστε να έχουμε την προσέγγιση bottom-up, εκ των κάτω προς τα άνω, ώστε να έχουμε μια προοπτική σε σχέση με την top-down από πάνω προς τα κάτω ανάπτυξη με ένα κατάλογο προτεραιοτήτων για τα σχέδια αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περίοδος για αυτά τα προγράμματα που αποσαφηνίστηκε όχι από μια καθορισμένη ημερομηνία του ημερολογίου αλλά από τότε που θα αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός Πρόκειται εδώ και για θέματα επίγοντα που πρέπει να προαθούν για την διαφάνεια και την ασφάλεια των επενδύσεων και τη χρηστή διαχείριση. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, σε αυτά δόθηκε μεγάλη σημασία στην, ε, στην επιμέρους ε, ε, ανάγκη ανταπόκρισης ε, στις ξεχωριστές ανάγκες των περιοχών και περιφερειών. Με ανάλυση των κριτηρίων κόστους κόστους-οφέλους. προτάθηκε ένας διαπραγματευτικός μηχανισμός ώστε να μην υπάρχει μονομερής επιβολή από κάποιο κράτος μέλος σε σχέση με το κοινό αυτό κοινοτικό εγχείρημα ένας μηχανισμός που είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν με λογικά, με θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την αδειοποίηση, την χωρίση αδειών, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ε, οργανισμού one stop shop και σε μία περίοδο τριών ετών πρέπει να ε, τύχουν ε, υπεράσπισης. Επιδοκιμάζουμε η περίοδος για αυτά τα τρία χρόνια με θετικά κίνητρα και ε, όσον αφορά την εφαρμογή του One Stop Shop, της ε, μίας θηρίδας ε, και της υποχρέωσης να υπάρχει παρακολούθηση της εφαρμογής με κίνητρα και έπαθλα για τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την υλοποίηση και την εποπτεία, ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών παρόχων στα διαφορετικά κράτη-μέλη, ώστε να έχουμε fast first movers με κίνητρα, κίνητρα που πρέπει να τους δώσει τη δυνατότητα να κινηθούν ταχύτερα. Αντί να υπάρχουν ε, αντικίνητρα ή πρόστιμα ή κυρώσεις σε σχέση με την ε, υλοποίηση της ε, ε προσέγγισης αυτής ε, για τους στόχους της διασύνδεσης. Όπως ξέρουμε οι στόχοι της, για τη διασύνδεση καθυστερούν ελήφθησαν μέτρα για να υποχρεωθούν οι πάροχοι των σχεδίων αυτών να υλοποιήσουν τα όσα υποχρεούνται έγκαιρα και σε σχέση και ε, με τις σαφείς ε, προθεσμίες ε, για να μπορούν να γίνουν δεκτά από τους εταίρους αυτά για την αδειοποίηση των προγραμμάτων να υπάρχει μια εναλλακτική λύση όσον αφορά την ε, ταχεία εφαρμογή. Μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει, υπάρχει η πρόταση συντονισμού για την συνεργασία και προαγωγή του συστήματος. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Systems coordination. Δηλαδή, σε σχέση με τον συντονισμό θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια του δικτύου για να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι blackout που ε, θα είναι πιθανότερη λόγω του ε, σύνθετου περίπλοκου χαρακτήρα του δικτύου θα πρέπει να γίνεται χρήση και εκμετάλλευση των υποδομών ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα δίκτυα του στο μέλλον. Δεν προτείνουμε ένα νέο οργανισμό ή φορέα. Θέλουμε να υποβάλλονται οι προτάσεις ε, με βάση το τι γίνεται μέχρι σήμερα όπως και στο παρελθόν και να υποβάλλονται οι προτάσεις τους με βάση αυτούς τους στόχους. Όσον αφορά την χρηματοδότηση, δημόσια χρηματοδότηση, είναι σημαντικό να αποφύγουμε στρεβλώσεις στην αγορά και ε, να μπορέσουμε να δράσουμε, αλλά σε σχέση όσον αφορά με ειδικέ δράσεις για μη εμπορικά ε, κερδοφόρα σχέδια. Η πρόταση είναι ότι έχουμε σύνολο, σύνολο μέτρων που όμως ε, δεν υπάρχει και η απόλυτη βούληση, η θετική βούληση των κρατών μελών για να προαχθούν. Χρειάζεται αυτή η κοινή βούληση για τα ε, κοινά αυτά σχέδια, για την αδειοποίηση και τις προθεσμίες ε, που θα λειτουργήσουν ώστε να είμαστε υπέρ της πρόοδου που θα μπορέσει να επιτευχθεί. Μέχρι σήμερα είμαστε πολύ βραδείς και καθυστερημένοι, καθυστερούσαμε πολύ. Θα πρέπει εδώ σε σχέση με την εθνική διατήρηση ε, κάποιων εξουσιών να μην αποδυναμωθούν αυτές οι προτάσεις. Θα είναι σημαντικό λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να έχει στη διαπραγμάτευση που προσεγγίζει μια ενωμένη φωνή, ενωμένη φωνή που θα είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της πρότασης της Επιτροπής για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Αγοράς και για μια πρόταση που είναι αναγκαία να έχουμε αποτελέσματα πανευρωπαϊκά και όχι μόνο εκεί όπου υπάρχει απόλυτη συνένεση για την διεύρυνση του δικτύου. Ευχαριστώ τον, τους κοιόδης εισηγητές για τις ανταλλαγές απόψεων και έχω την ελπίδα, ευελπιστώ ότι η συνεργασία αυτή θα διασφαλιστεί και θα διατηρηθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ για τη συνεργασία όσον αφορά και όλους που συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν οι σκεώδεις εισηγητές, ο κύριος Σαρδάργας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρεί, συγχαρώ τον εισηγητή για την φιλόδοξη πράγματι αυτήν έκθεση. Και εγώ συμφωνώ με τη γενική άποψη του εισηγητή που θεωρεί αυτό το κανονισμό επίκαιρο, σημαντικό και πολύ καλογραμμένο. Τον συγχαίρω ακόμη μια φορά γιατί έλαβε το θάρρος μάλιστα και να βελτιώσει την πρόταση. Υποστηρίζω τις κύριες γραμμές και στρατηγική του να ενδυναμωθεί δηλαδή η θέση της Ένωσης Ας μην επαναλάβω πόσο εκτιμώ το α ή το β μέρος του κανονισμού, της έκθεσης και των τροπολογιών. Απλώς θα πω ότι γενικά υποστηρίζω τις κύριες γραμμές. Τώρα θα επικεντρωθώ στα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε συμβιβασμούς. και φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί πολύ και η θέση του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο. Πρώτον, τα προβλήματα δεν είναι στρατηγικής ή γενικής φύσεως. Πρόκειται για τεχνικά λεπτομέρειες. Και το κύριο διαδικαστικό πρόβλημα είναι η ταύτιση του ορισμός του προγράμματος κοινού ενδιαφέροντος. Ο εισηγητής δεν άλλαξε αλλά επαναδιατύπωσε την διαδικασία, αυτή η διαδικασία είναι τώρα. Εγώ υποστηρίζω μερικά από αυτά που λέει, αλλά θα τροπολογήσουμε κιόλα. Γιατί έχουμε και εμείς μερικές διαφορούλες. Μία από αυτές είναι ότι στον κανονισμό αυτόν προβλέπεται μια πρόταση ταύτισης κανονισμο αυτων προβλεπεται κοινού ενδιαφέροντος επιλογής τους δηλαδή αυτών των ΠΚΕ και χωρίς καμία ιεράρχηση ή διαφοροποίηση ασαφώς γίνεται λόγος. για το ότι μάλλον οι κομισιόν ή ορισμένες επιτροπές πρέπει να κάνουν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει το πράγμα σαφέστερο η κομισιόν να κάνει την επιλογή. Και βέβαια θα δούμε, θα φροντίσουμε να, φροντίσουμε, να φροντίσουμε να διορθώσουμε και τη διατύπωση. Άλλα στοιχεία που δεν μπορώ να δεχτώ Λεπτομέρειες είναι και αυτά, αλλά έχουν κάποιο νόημα. Η αναφορά στους στόχους αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών δεν δικαιολογούνται παρά μόνο στη γενική εισαγωγή, στο σκεπτικό, αναφορά στους στόχους 2020 κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να τα γράφουμε αυτά και μέσα στη ίδια τη διαδικασία επιλογής των ΠΚΕ. Είναι υπερβολική η λεπτομέρεια γιατί η όλη στρατηγική αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Δεν πρέπει να τα βάζουμε εκεί αυτά. Τώρα, η δημιουργία των περιφερειακών ομάδων ή ο ορισμός τους, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό πρέπει να προσέξουμε πολύ αν θα τις επεκτείνουμε τις ομάδες αυτές ή όχι. Ίσως να πούμε ότι σε άλλα κείμενα πρέπει να διευθετηθούν αυτά. Αλλά η ευρύτερη αλλα κειμενα πρεπει να διευθυντηθουν αυτα χρηστών και χρηστριών, παραγωγών κλπ. για να είναι πιο διαφανής αυτή η διαδικασία να υπάρξει κάποια διαβούλευση. Μπορούμε να το γράψουμε, αλλά για κανονική συμπερίληψη δεν νομίζω ότι πρέπει να αποκλειστεί. Αυτά νομίζω ότι μπορεί και να αρκούν. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο, γιατί αλλιώς ε, δεν θα καταφέρουμε να τελειώνουμε. Η κυρία Βάλεν. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Ντεκάμπος για την εξαιρετική του έκθεση. Και υπάρχει εδώ και υποστήριξη το, σε σχέση με την, τους εμπλεκόμενους τους υποδομές. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η έκθεση αλλά και σε σχέση με το θέμα της εισήγησης για τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών χωρών. Είχαμε και ακρόαση σήμερα το πρωί που μας δείχνει ότι έχουμε τεράστιο, ένα τεράστιο πελώριο μηχανισμό ευρωπαϊκό σε σχέση με αυτά. Είναι ένα επαναστατικό μέσο αυτό σε πολλές πτυχές διοικητικά, οικονομικά, χρηματοδοτικά. Πολλές προκλήσεις εδώ συγκλίνουν που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μία από αυτές τις προκλήσεις για μας τουλάχιστον είναι να αποφύγουμε την ανάμιξη στην αγορά και την δημιουργία μη ίσου πεδίου δραστηριοποίησης στον ανταγωνισμό ιδιαίτερα όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα και τηλεπικοινωνίες. Μια από τις προτεραιότητες σε αυτόν το, σε αυτό τον κανονισμό θα είναι τα κριτήρια για την εκπόνηση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ολοκλήρωση στην αγορά και την πρόθεση του ανταγωνισμού, αποφεύγοντας στρεβλώσεις, ώστε να μην έχουμε ε, την ε, στρέβλωση σε σχέση με, κάποιες, ε, με κάποια σχέδια. Δεν είναι δυνατόν μόνο τους διαδρόμους να εξετάσουμε, αλλά και τις εθνικές υποδομές, ώστε να υπάρχει αναγκαία διασύνδεση το θέμα της αδειοδότησης είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο να υπάρχουν απλουστευμένες ε, αποτελεσματικές διαδικασίες στο εθνικό επίπεδο εκάστοτε που έχουν, τεράστια σημασία. Συμπεριλαμβάνω αυτό στην έκθεσή μου σε σχέση με κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, σκεπτικών ή εδαφείων. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις για αυτή την έκθεση. Πρώτα, η PCI, η επιλογή PCI προγραμμάτων σχεδίων κοινού συμφέροντος έχει κέρια σημασία και ενώ εργαζόμαστε σε σχέση με την υπόθεση εργασίας ότι ο εισηγητής άνοιξε αυτή την άκαμπτη διαδικασία και την καθιστά πιο απελευθερωμένη, πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Χρειάζεται αποτελεσματικότητα οπωσδήποτε. Το γεγονός ότι κύριος ρόλος δίνεται στις ε, DSOs είναι κάτι αμφισβητήσιμο μια και δεν έχουν μια πλήρη εικόνα αυτών των δικτύων. Οι, ε, ε, όσοι εκμεταλλεύονται τα δίκτυα αλλά και οι χρήστες πρέπει να έχουν ρόλο και λέγει στο, στα όσα θα μεταξελιχθούν σε σχέση με τις ε, τοπικές αγορές ε, και την πιο αποτελεσματική προσέγγιση σε σχέση με κόστος-όφελος. Για τα ενεργειακά θέματα θα είναι παράλογο, για παράδειγμα, να μην ε, ενταχθούν στον κατάλογο αυτά τα σχέδια τα οποία υποστηρίζονται από τους ε, ιδιώτες επενδυτές αλλά δεν υποστηρίζονται από τις TSOs. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας ε, στην επιλογή, όμως ε, η διαχείριση είναι ένα θέμα μαύρου κουτιού. Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, πώς θα λαμβάνονται αποφάσεις σε τέτοιες ομάδες. Είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα, να εμβαθύνουμε σε αυτό. Άλλο θέμα αυτό το οποίο αφορά την αρχιτεκτονική για τον κατάλογο PCI και την μεθοδολογία που υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προτάσεις του εισηγητή. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που δεν θα είναι βιώσιμος, που θα οδηγεί σε οπωσδήποτε επικαλύψεις ε, και αναποτελεσματικότητα για τον πρώτο κατάλογο σε σχέση με τον Ιούλιο 2013 που ακούσαμε ότι εργάζεται επ' αυτού ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότι αυτή η πρόταση ακόμα δεν έχει εγκριθεί τι θα γίνει. Θα πρέπει να έχουμε μια μεταβατική περίοδο καλύτερα, ώστε σε σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα να ανταποκρίνονται στις ε, προδιαγραφές και στα κριτήρια, ώστε να, υπάρχει ίση να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα σχέδια για την ε, ασφάλεια το, της τροφοδότησης και των ενεργειακών ε, αγανών των αναγκών αυτών πρέπει να συμπεριληφθούν και τα θέματα αποθήκευσης ε, και τα θέματα τροφοδότησης. Έχω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις, αλλά αυτές μεταξύ μου και εισηγητού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τον εισηγητή για την ποιότητα της έκθεσής του και τη συνεργασία που είχε με όλους τους κοιόδης. Για μας Υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία στην έκθεση αυτή, ιδιαίτερα το ότι μας εξήγησε και τα θέματα του λεγόμενου έξυπνου δικτύου κλπ. Γιατί καμιά φορά μιλάμε μόνο για τους αυτοκινητοδρόμους της επικοινωνίας και λιγότερο για την εξοικονόμηση ενεργείας που για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης στηρίζουμε τον εισηγητή ναι την πρόταση που μας κάνει για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΡ για να δοθούν ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές Τρία θέματα τώρα επί των οποίων θα θέλαμε να επιμείνουμε. Πρώτον, οι υποδομές του ηλεκτρισμού. Η κατανομή είναι δύο τρίτα ηλεκτρισμός, ένα τρίτο αέριο. και σε αυτό επιμένουμε. Επίσης, η παρουσία στο κείμενο αυτό του ΣΥΣΕΣ μας φαίνεται κάπως άχρηστη. Γιατί εδώ μιλάμε για κείμενο που πρέπει να λύσει τρία προβλήματα. Τη χρήση των ανανεωσίμων, την αγορά ενεργείας και την ασφάλεια προμηθειών ενεργειακών. Το CCS δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από τα τρία. Μιλάει για την προοπτική του 2020 και ξέρουμε ότι μέχρι τότε δεν θα έχει εμπορικές προοπτικές το CCS. Ακόμα πειραματικό είναι. Και δεν βλέπουμε λοιπόν γιατί να βάλουμε αυτή την παραπομπή εδώ. Δεύτερον, το θέμα της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής επιλεξιμότητας των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος ή και. Εμείς θέλουμε να διευρυνθούν οι περιφερειακές ομάδες. Όσες είναι δραστήριες και ενεργές, δηλαδή και τους καταναλωτές και καταναλώτριες και τις ομάδες που ούτως ή άλλως θα παρέμβουν στη διαδικασία. Αν θέλουμε, όπως θέλουμε εμείς, να υπάρξει και ταχύτητα στην κατασκευή αυτών των υποδομών, τότε πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία επέκτασης αυτών των ομάδων για να υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή τους. Ε, και αυτό αφορά επίσης την μεθοδολογία την ανάλυση κόστους οφέλους. Στην ανάλυση αυτή κόστους οφέλους και μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα, δεν μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα για οδική χάρτα μέχρι το 2020 και να παραλείπουμε σε αυτές τις αναλύσεις τους στόχους, συνεργειακούς στόχους που θέτει στον εαυτό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, τρίτον, να μην βάλουμε σε αντιπαράθεση τη συμμετοχή του κοινού με την αποτελεσματικότητα ούτε την οικονομία με την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε να συνδυαστούν αυτά. Διαβούλευση του κοινού, προστασία του περιβάλλοντος, διότι το να λέμε ότι θα τα λύσουμε όλα σε τρία χρόνια μας φαίνεται λάθος. Αν δεν τα καταφέρουμε σε τρία χρόνια, μπορεί να χαθούν μερικά σχέδια αντί να τους δοθεί ο χρόνος που απαιτείται για να εφαρμοστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, να συγχαρώ τον συνάδελφο Αντώνιο Κορέλια, ο οποίος εργάζεται αποτελεσματικότατα. Και σέβεται και ιδιαίτερα τη συνεισφορά των σκεωδών εισηγητών. Εγώ για μία ακόμη φορά θα ήθελα να τονίσω στον εισηγητή μερικά από τα σημεία που θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά σε αυτόν τον κανονισμό. Πρώτο, θα πρέπει να ενισχύσουμε ένα σχεδιασμό με ευρωπαϊκό όραμα. Αυτό είναι το, ε, το το, κουσούρι που είχε μέχρι σήμερα η ενεργειακή πολιτική και πρέπει να το αποφύγουμε. Ξεπερνώντας δηλαδή την το, εθνικό όραμα για την αναδιάρθρωση των υποδομών. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα εθνικά συμφέροντα και να καταφέρουμε να, να απεικονίσουμε ένα σχέδιο ευρωπαϊκής εμβέλειας. Εμείς θα είμαστε πάντα υπέρ της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών ε, θεσμών και πιο συγκεκριμένα της Κομισιόν. Σχετικά με τις περιφερειακές ομάδες, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Και αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα στους κανόνες λειτουργίας αυτών των περιφερειακών ομάδων και πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο και στο σύστημα έγκρισης συμφωνιών. Πρόκειται για ένα σημείο πολύ σημαντικό για την ε, ανάπτυξη και εξέλιξη των σχεδίων και δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Τέταρτο, θέλω να σταθώ στην ανάγκη του να τονίσουμε ότι οι υποδομές οι οποίες δεν έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα αλλά είναι απαραίτητες για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και βοηθούν στην ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών δεν θα πρέπει να υποστούν διακρίσεις κατά τη στιγμή της επιλογής των σχεδίων ευρωπαϊκού συμφέροντος. Ευρωπαϊκό συμφέρον δεν είναι μόνο τα διασυνοριακά σχέδια. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν εθνικά σχέδια, μη διασυνοριακά, τα οποία όμως έχουν ευρωπαϊκή σημασία. Πέμπτο, θέλω να υπογραμμίσω την πολιτική συνοχής μεταξύ των ενεργειακών πολιτικών και των άλλων πολιτικών. Εδώ θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι άλλοι συνάδελφοι προηγουμένως. Η συνεκτικότητα, η συνάφεια των πολιτικών είναι πολύ σημαντική. Η πολιτική για το κλίμα, πολιτική των μεταφορών, βιομηχανική πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική. Όλα αυτά είναι βασικά εάν θέλουμε να έχουμε ένα συνολικό, ένα πλήρες όραμα και ευρωπαϊκές εμπνεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι η καλύτερη υποδομή είναι αυτή που δεν χρειαζόμαστε. Και η έμφαση στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα πάντα θα είναι λίγη. Εγώ Ίσως ε, να είμαι εθεροβάμων ε, και θέλω να κατεβάσουμε τα τρία χρόνια στα δύο. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, όπως επίσης ε, και την ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών. Ευχαριστώ. συνάδελφος Γιούρουκ. Ευχαριστώ. Και συνεχίζοντας και εγώ αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι μια πολύ ισόρροπη έκθεση και σε σχέση και με την πρόταση της Επιτροπής που ήταν καλή κατάφερε να βελτιώσει τα πράγματα ο εισηγητής. Τρεις παρατηρήσεις έχω σε σχέση με την πρόταση. Η πρώτη παρατήρηση. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Ένα ως μηδενικό σημείο Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις υφιστάμενες υποδομές προτού αναπτύξουμε καινούριε. Πολλά πρέπει να κάνουμε στις μεταφορές σε σχέση με υφιστάμενες ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας καλύτερη χρήση των υποδομών που υφίστανται και αποφεύγοντας έτσι δαπανηρές εξελίξεις νέων υποδομών. Κάθε φορά όταν συζητούμε για επενδύσεις σε νέες υποδομές, πρέπει να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε πώς χρησιμοποιούμε τις υφιστάμενες υποδομές. Σε μια περίοδο κρίσης αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Προτείνω τώρα το εξής. Αξιολόγηση κριτηρίων, ανάλυση κόστους ωφέλους, όπως προτείνονται. Πρέπει να έχουμε δομημένα, διαρθρωμένα <clears throat> πρότυπα κριτήρια για όλα αυτά. Αυτό δείχνει ότι θα υποστηρίζουμε μόνο τα πιο σημαντικά προγράμματα που θα είναι προτεραιότητας προγράμματα. Τρίτη παρατήρηση, θα μακρηγορήσω λίγο περισσότερο, θα χρονοβορήσω σε αυτή την παρατήρησή μου. Έχουμε κάποια πιο περίπλοκα ζητήματα όσον αφορά λεπτομέρειες, όσον αφορά περίπλοκες εκθέσεις, όπως έχουμε αυτή την έκθεση ενώπιόν μας τώρα. Βλέπω και βρίσκω προβλήματα όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, όπως εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, στο δεκαετές πρόγραμμα. Ένα, σημείο προβληματισμού και οι περιφερειακές ομάδες ή ε, περιφερειακές οργαν... περιφερειακοί οργανισμοί. Αντιφατικά εδώ κάποια πράγματα. Το άρθρο 3 σημείο 7 ήταν αντιφατικό. Προτείνει η περιφερειακες περιφερειακοι οργανισμοι αντιφατικα εδω καποια πραγματα το αρθρο Επιτροπή οι περιφερειακές αυτές οργανώσεις ή ομάδες να υποβάλουν προτάσεις επενδυτικές προτάσεις και Και με έγκριση και υποστήριξη των, της ε, Ευρώπης, ευρωπαϊκή υποστήριξη θα εντάσσονται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Αν δούμε όμως το NSP βλέπουμε το αντίθετο ακριβώς να γίνεται. Μόνο επενδύσεις καλύπτονται. Μόνο εκείνες οι επενδύσεις θα μπορούν να θεωρούνται όπως, ως επενδύσεις προτεραιότητας εκείνες που θα έχουν ήδη ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα θα με ικανοποιούσε ιδιαίτερα αν μπορούσε να αποσαφηνίσει αυτή την αντίφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιφατικότητα εδώ. Με τις τροπολογίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά πρέπει να γίνει και παραπέρα δουλειά. Νομίζω η πρώτη ε, διατύπωση είναι η σωστότερη. Οι περιφερειακές ομάδες ή οργανισμοί θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τέτοιες προτάσεις. Ποιος όμως θα κάνει την ανάλυση ωφέλους σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτή η πρώτη προσέγγιση είναι η ορθότερη πιστεύω. Διότι αν οδηγηθούμε στο παράτημα 3, εκεί μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο σε προγράμματα που έχουν ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα. Τώρα, θα αποδυναμωνόταν το συνολικό πακέτο και θα αποδυναμωνόντουσαν και οι περιφερειακές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει λοιπόν, λοιπόν να αποσαφινιστεί αυτή η αντίφαση και να αρθεί ευχαριστώ. κυρία Βαμπρέντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Θα ήθελα Να αναφέρω ότι πρόκειται για μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική σε αυτή τη φάση που η Ευρώπη δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον για την ενέργεια. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όπως και οι εθνικές αρχές νομίζω ότι θα πρέπει να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο κυρίως ε, για την τιμολόγηση στον καταναλωτή. Πρέπει να ορίσουμε τους στόχους μας μακροπρόθεσμα, τι θέλουμε μέχρι το 2050, πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία και θα πρέπει να βασιστούμε 100% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να ανανεώσουμε το ε, δίκτυο, το ηλεκτρικό δίκτυο από σήμερα. 200 εκατομμύρια ε, αναφέρει η Κομισιόν, 60 εκατομμύρια για το φυσικό αέριο. Εγώ νομίζω ότι μακροπρόθεσμα το δίκτυο θα πρέπει να εξαρτάται απόλυτα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να δούμε επίσης τις προπτικές του 2030-2050. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει τι γίνεται με τα τοπικά κέντρα διανομής και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ η κυρία Ντελκαστίγιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα είμαι εγώ η τελευταία, γιατί θα μιλήσουν κι άλλοι. Και μίλησαν κι άλλοι πριν από μένα, θα συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή με εξαιρετικό τρόπο, επαγγελματικότητα, πραγματικά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να, να, πω ότι θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για τις τροπολογίες που εισηγαγε νέες παραγράφους, τροπολογία 62 στο άρθρο 13 στη δεύτερη παράγραφο και στην τροπολογία 63 στο άρθρο 13, μια δεύτερη παράγραφο β. Αυτό το, η δημιουργία ενός συστήματος benchmarking για το κόστος των επενδύσεων για τις διασυνοριακές συνδέσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι πολλές φορές οι επενδύσεις σε δύο μεριές των συνόρων, πολλές φορές σε, τρεις, σε τρία διαφορετικά σύνορα, οδηγούν σε μία στασιμότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η θέση του εισηγητή και μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα. Τώρα, για τις περιφερειακές ομάδες είναι δύσκολο να ορίσουμε τις ε, περιφερειακές ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες ευκαιρίες έχουν για να μπορέσουν να περάσουν αυτά τα σχέδια. Ε, ο διαδρομος βορράς, ε, βορρά-νότου για τον ηλεκτρισμό θα μπορούσαμε να έχουμε δύο υποδιαδρόμους. Από το νότο στο κέντρο, Southwest και Central West. Αυτά θα έπρεπε να τα συζητήσουμε και μετά τα υφή δίκτυα. Έχουμε ένα σωρό αναφορές στην έκθεση της Επιτροπής, αλλά θα έπρεπε να ενισχύσουμε με ποιο κριτήριο θα χρηματοδοτήσουμε τα smart grids, τα εφή δίκτυα. Θα πρέπει να έχουμε έναν ειδικό κανονισμό που θα εξετάζει μόνο το θέμα των smart grids, γιατί αλλιώς αυτό το σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων θα παραμείνει ένα χολό σχέδιο. Κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Και εγώ τον εισηγητή. Ιδιαίτερα για την τροπολογία 1, διότι είναι ουσιώδες να μην ξεχνάμε τη σημασία της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας να μιλάμε για υποδομές. Κομισιόν θεωρεί ότι αν καταλήξουμε στο 20% βελτίωση το 2020, αυτό θα σημαίνει εξοικονόμηση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Πράγμα που μπορούμε να το δαπανίσουμε μετά για την παραγωγή και διανομή ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στις υποδομές, αλλά επίσης σημαντικότατο είναι να μην χρειάζεται να επενδύσουμε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Γι' αυτό μου άρεσε πολύ αυτή η τροπολογία. Τώρα, για, το υπόλοιπο, για την κατανομή των ε, επενδύσεων μεταξύ αερίου και ηλεκτρισμού. Πρέπει να σκεφτούμε στρατηγικός πώς. Δηλαδή, η απανθρακοποίηση της οικονομίας θα εξαρτηθεί από την οικονομία, από τον ηλεκτρισμό για τις μεταφορές, για τη θέρμανση και γι' αυτό θα ήθελα να δοθούν περισσότερα χρήματα για τον ηλεκτρισμό, τα δύο τρίτα ας πούμε, παραπάνω από τα δύο τρίτα μάλλον. Δεν έχω καμία αντίρρηση για την αποθήκευση του διοξιδίου, αλλά δεν νομίζω ότι σχετίζεται με αυτήν την πρόταση που αφορά το τι θα κάνουμε πριν το 2020. Ακόμα το εξετάζουμε το θέμα της αποθηκεύσεως. Δεν πρόκειται μέχρι το 20 να έχει εφαρμοστεί εμπορικά. Τρίτον, όσον αφορά τις διαβουλεύσεις είναι πολύ σημαντικό να είναι τεχνολογικός ουδέτερες. Γιατί ένας λόγος των καθυστερήσεων στα, στην έγκριση των προγραμμάτων υποδομών είναι ότι μερικοί αντιδρούν σε μία πτυχή όπως ας πούμε τα σύρματα και δεν βλέπουν το σύνολο και το ίδιο ισχύει και για τις αναλύσεις κόστους-οφέλους. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Γιατί εντάξει μπορούν τμήματα των σειρμάτων να θάπτονται. Αλλά μπορεί αυτό να κοστίζει περισσότερο. Αν το πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί νωρίτερα θα μπορούσε να εγκριθεί χωρίς το θάψιμον. Πρέπει να τα όλα αυτά υπόψη μας στις αναλύσεις κόστους και ωφέλους. Αυτό εννοώ τεχνολογικό σου ουδέτερη ανάλυση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Βιδάλ Κουάδρας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση του συναδέλφου Κορέα η Κάμπος διέπεται από μια γενική αντίληψη την οποία συμμεριζόμαστε όλοι σε αυτήν την Επιτροπή. Πρόκειται για την κεντρική ιδέα ότι μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας δεν είναι εφικτή άμα δεν έχουμε μία φυσική υποδομή που επιτρέπει την υλοποίησή του. Και μέσα από αυτήν την αδιαμφισβήτητη διαπίστωση η έκθεση του συναδέλφου τίνει προς μία αυθεντικά ευρωπαϊκή κατεύθυνση που του αξίζει συγχαρητήρια. Εμείς καταβάλαμε προσπάθειες για να υπά... εδώ και χρόνια για να υπάρξει αυτή η ενιαία αγορά. Αλλά υπάρχουν κυβερνήσεις που σέρνουν τα ποδάρια τους και άλλοι που κολλησουργούν. Πρέπει με αυτή την έκθεση να κάνουμε ένα άλλο βήμα προς τα μπρος για, τη λύση που οι περισσότεροι σε αυτήν την Επιτροπή επιθυμούν. Χρειάζεται πρόβλεψη μιας διαδικασίας σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αρνηθεί ένα σχέδιο κοινού συμφέροντος σε μία, ε, στην επικράτειά του, ούτως ώστε να, μπορούμε, ούτως ώστε να μην έχουμε εμπόδια. Επίσης, δείκτες για τον υπολογισμό του κόστου στα διά... των επενδύσεων στα διάφορα κράτη-μέλη διότι αυτό προσδίδει διαφάνεια και περιορίζει τους εξυπνάκηδες. Επίσης, σχέδια πρέπει να ληφθούν υπόψη σχέδια τα οποία στο παρελθόν είχαν θεωρηθεί σχέδια ε, ευρωπαϊκού συμφέροντος. Δεν θα ήθελα να ξεχάσω να αναφέρω ευνοϊκά την ανάγκη διπολικών ροών που αναφέρει ο εισηγητής Επίσης ότι οι τερματικοί θα πρέπει να αποτελούν τμήμα των υποδομών και επιμένω θα πρέπει να τελειώνουμε με τις ενεργειακές νησίδες. Οι εγκαταστάσεις ε, ε, ενεργειακής αποθήκευσης με υδραυλικές αντλίες ε, δεν μπορούν να, να δεν μπορούν να τις διαχειρίζονται τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Θέλω ξανά να συγχαρώ τον Κορέα Κάμπος, μετά από την έκθεσή του θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της συναδέλφου Ριέρα που δεν είναι παρούσα. Και θέλω να υποστηρίξω την έκθεση του εισηγητή Αντώνιο Κορέια Δεκάμπος. Εξαιρετική δουλειά, το είπαμε. Δεν θέλω να επιμείνω. Η έκθεση κλαμβάνει σωστά την προβληματική τη έλλειψης κοινών υποδομών μεταξύ των διαφόρων χωρών και για τη διαχείριση αλλά και για τη δημιουργία μιας κοινή ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Στην τωρινή φάση κρίσης αυτό το πλαίσιο δυσκολεύει ιδιαίτερα τη λήψη απόφασης για επενδύσεις. Πράγμα που υποχρεώνει να τους καταναλωτές να υπόκεινται το βάρος των επενδύσεων στον τομέα αυτό. Και η σύγκριση κόστους που αναφέρει ο εισηγητής είναι μια πολύ χρήσιμη αναφορά για να, βελτιώ, για να διασφαλίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Όλα αυτά θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία των συμφερόντων της βιομηχανίας και των καταναλωτών στόχοι πολύ σημαντικοί για την Επιτροπή μας. Ένα άλλο θέμα είναι η υποδιέρεση των, διαδρόμων για τον ηλεκτρισμό. Έτσι όπως είναι σήμερα, δύσκολα μπορεί κανείς να τους διαχειριστεί. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε τις υποδομές των περιφερειακών δικτύων που έχουν ήδη την εμπειρία λειτουργίας. Συνάδελφος Τούρμες. Ε, ε, Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Εγώ τώρα εξετάζω το Connecting Europe Facility και όπως είπαν μερικοί δίνεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για τον ηλεκτρισμό χωρίς να αγνοούμε και το αέριο αλλά όπου χρειάζονται λιγότερες επενδύσεις κυρίως στις ηλεκτρικές υποδομές. Δεύτερον, πριν από δύο-τρία χρόνια έμαθα κάτι ότι ανακάλυψα το εξής. Τα προγράμματα υποδομών που τελικά καταλήγουν να παράγουν ηλεκτρισμό από το κάρβουνο μπορεί να επανεισάγονται στην ε, Ευρωπαϊκή Αγορά Ενεργείας Ουκρανία, Σερβία, Ρωσία και ίσως στην Ισία, Ιταλία παράγουν από το κάρβουνο ηλεκτρισμό και μεταδίδεται από ένα σύρμα καλώδιο στην Ένωση και άρα δεν υποβάλλεται στα δικά μας κριτήρια. Αυτό δεν είναι το ίσιο γήπεδο που λέγαμε. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό γιατί Μπορεί και 10.000 ΜΒ να καταναλώνονται έτσι με τέτοιο τρόπο. Πρέπει να βρούμε μια λύση για αυτού του είδους τον ηλεκτρισμό. Τέλος μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη μπορούμε να δεχτούμε τότε έναν προϋπολογισμό βάσει βάση του οποίου οι αποζημιώσεις που δίνονται στους διαχειριστές των δικτύων είναι τόσο μικρές όσο σήμερα. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει κάτι παράλογο. Γιατί μειώσαμε δραστικά τον προϋπολογισμό ενώ παράλληλα ζητάμε από τους διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων να συνεργάζονται όλο και περισσότερο. Αυτό είναι λογικό, πρέπει να το δούμε και αυτό και είναι καλή ευκαιρία η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Θέλω να προσθέσω τη φωνή μου σε εκείνους που συνεχάρισαν τον εισηγητή για μια πολύ καλή έκθεση. Με ιδιαίτερη χαρά <clears throat> παρακολουθώ και ακούω τις θέσεις των μελών αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και νομίζω όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η πρότασή μας την χάνει μεγάλη υποστήριξη και ότι γίνονται κατανοητές οι αρετές της, διότι είναι σωστό, είναι μια επαναστατική πρόταση. Για μια πρώτη φορά έχουμε μια πραγματικά αυθεντικά ευρωπαϊκή προοπτική για τα θέματα ηλεκτρικής ενέργειας ρεύματος και φυσικού αερίου στις υποδομές. Πολύ ενθαρρυντικό είναι αυτό. Και για το εύρος, το φάσμα αυτό, πιστεύω ότι φυσικά έχουμε πολλαπλά θέματα υποδομών, δίκτυα διανομής, αγωγούς, αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου, ε, αποθήκευση αερίου έχουμε και θέματα που ίσως πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και να επανεξεταστούν γιατί είναι μια πολύ ανταγωνιστική αγορά αυτή και στρέβλωση στις αγορές είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε και αυτό αναφέρθηκε σε σχέση με τα όρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις συζητήσεις. Διάβασα για το CCS. Αν θέλουμε να έχει κάποια ευκαιρία, καλό είναι να δείξουμε τι ποιες ανάγκες υπάρχουν σε σχέση για τα θέματα διοξιδί του άνθρακα. Πρέπει αμέσως να ξεκινήσουμε με μια ευρωπαϊκή προοπτική σε, σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και το 2020 ως στόχο καταληκτικό που έχουμε και πρέπει να πετύχουμε αυτό το στόχο. Για τις περιφερειακές ομάδες ή οργανώσεις είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στις περιφερειακές αυτές ομάδες Εκεί υπάρχει κύριος ρόλος ε, για εκείνους ε, που προωθούν αυτά τα δίκτυα, τις ρυθμιστικές αρχές και τα κράτη-μέλη. Να σας υπενθυμίσω απλά ότι στη συνθήκη τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε θέματα υποδομών στην επικράτειά τους. Και πάλι, με άλλα λόγια, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν φυσικά όλα αυτά. Και έχουμε και την τροπολογία 63 που σίγουρα θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τα κράτη-μέλη για το θέμα της, διότι αν δεν δέχονται τα κράτη-μέλη θέματα υποδομών και θα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι πολύ προκλητικό, ιδιαίτερη πρόκληση για μας. Πρέπει πραγματικά να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία στις σχέσεις αυτές ταυτοποιώντας τα προγράμματα αυτά, τα σχέδια κοινού συμφέροντος προ όφελο του ευρωπαϊκού συμφέροντο που είναι το ζήτημα. Συμφωνούμε λοιπόν για την ανάγκη διαφάνεια. Συμφωνούμε να υπάρχει μια σαφή διαδικασία διεργασία λήψεων αποφάσεων. Σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν θα πρέπει όμως να αναμένουμε ίσως υπερβολικά πολλά και υπό το πρίσμα των όσων ανέφερα για το ρόλο των κρατών μελών. Όλα αυτά θα βοηθήσουν βέβαια, πιστεύω. Και είδαμε πολλές παρεμβάσεις ε, σε σχέση με την πρόταση αυτή ώστε να μπορέσει να προωθεί η ε, διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης ε, προγραμμάτων και σχεδίων κοινού συμφέροντος. Και έχουμε και το θέμα της αποδοχής, αποδοχής από τα κράτη-μέλη. CBA, Cost Benefit Analysis, ανάλυση κόστους Οφέλους. Και αυτό θα διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο. Καλή πρόταση είναι να ενισχυθεί αυτή η συνιστόσα καλοδεχούμενοι. Και αυτό είναι φυσικά το κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία αυτή θα υφίσταται τέτοια ανάλυση και θα, θα πρέπει να επιτρέπεται στις περιφερειακές ομάδες να ε, ασκήσουν τις ε, δικές τους αρμοδιότητες. Για τις αδειοδοτήσεις και τις αρμόδιες αρχές τροπολογία 56 πρέπει πραγματικά να αξιολογήσουμε και να δούμε μπορεί αυτή η δουλειά να επιτευχθεί. Ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει. Δεν είμαστε απόλυτα πεισμένοι ίσως για όλα αυτά. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα να έχουμε το πρόγραμμα συντονισμού τροπολογίες 2 και 72. Και πάλι βρισκόμαστε καθοδόν να έχουμε μεγαλύτερο εναρμονισμό σε σχέση με τα συστήματα. Πάλι όμως πρέπει να προσέξουμε να μην επιβάλλουμε, να μην περιορίσουμε τους εμπλεκόμενους σε ένα σύστημα το οποίο δομείται, οικοδομείται αυτή τη στιγμή σε σχέση για παράδειγμα με τα όσα είχαμε στις πρώτες δύο εβδομάδες της εκκίνησης το Φεβρουάριο δεν θα μπορέσει με διατάγματα να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Πρέπει να εμπλακούν όλοι σε πλήρη βαθμό για να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι υπάρχει γενικότερα ικανοποίηση με τις τροπολογίες όπως προτείνονται από τον εισηγητή για τα συναφή θέματα και ευελπιστούμε ότι και σε σχέση με εσάς που θα καταθέσετε τέτοιες τροπολογίες ότι θα πορευθούμε προς την ευκταία κατεύθυνση που επιθυμούμε και εμείς να δημιουργηθεί μια αυθεντικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά όπου όλες οι διασυνδέσεις θα εξυπηρετούν τον ανταγωνισμό, την αηφορία και την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Αυτοί είναι οι τρεις κύριοι άξονες ως στόχοι που πρέπει να επιτύχουμε με τις υποδομές. Πλήρως συμμορφούμενοι και ευθυγραμμιζόμενοι με το πακέτο για τις αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία πληροφορία θέλω. Πόσο χρόνο θα μου διαθέσετε. Five minutes. That's enough. Okay, thank you. Πέντε λεπτά, πολύ καλά. Πολύ ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ ευχαριστώ κύριοι εισηγητέ, αγαπητοί συνάδελφοι και εκπρόσωπε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θερμά εξαιρετικά λόγια και επένου σα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την καλοσύνη σα και την ευγένειά σα με τον τρόπο που αντιμετωπίσατε την έκθεσή μου. Όμως ευχαριστώ κυρίως επίσης τις προτάσεις που υποβάλατε για τις προτάσεις σας. Θα πάρω με τη σειρά της παρουσίασης τα θέματα. Πρώτα, από πλευράς του συναδέλφου Τσαοντάργα και σε σχέση με τον σκιώδη συγητή ΕΛΚ, νομίζω ότι σε σχέση με ένα ασφάλμα που υπήρξε γιατί έγινε λόγος για κλάστερς στην ομαδοποίηση των προγραμμάτων επιλογής και ουσιαστικά τα κλάστερς δεν διαχωρίζονται. Θεματικά είναι διαφορετικά. Είναι μόνο τμήματα των, του πίνακα, του κάθε του καταλόγου. Νομίζω αυτή η αποσαφήνιση οφείλεται σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να γίνει. Σε σχέση με τις περιφερειακές ομάδες ή οργανώσεις, το δίλημα από πλευρά συναδέλφου Σαουντάρκας που θα ήθελε να επανέλθουμε στη διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ έχουμε το δίλημα για τη συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Είχαμε πολλά αιτήματα και πολλές πιέσεις που ασκήστηκαν από τους stakeholders, από τους εμπλεκόμενους να διευρυνθούν αυτές οι πτυχές. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι όλο και περισσότερο όταν διευρύνεται αυτό το πλαίσιο τόσο και πιο δύσκολη είναι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Και σε σχέση και με την τελική άποψη εξετάζοντας τις τροπολογίες στην οποία μπορούμε να καταλήξουμε. Συνάδελφε Βάλιαν που πιστεύετε ότι... Τι είπατε? Μάλιστα, που πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί φυσικά να αποφύγουμε τον δεσπόζοντα ρόλο κάποιων stakeholders. Συμφωνούμε απόλυτα. Η αλήθεια όμως είναι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο κυριότερος stakeholder, ο πάροχος, ο εκείνος που παρέχει και ε, παράγει αυτές τις υπηρεσίες είναι ο πιο σημαντικός και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό ως συνιστόσα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σαν να είχε εγκριθεί αυτή η πρόταση αναφέρθηκε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό και το ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βιάζεται λέει υπερβολικά. Για αυτούς όλους τους λόγους εμείς τι κάνουμε. Θέλουμε τα τρία χρόνια να μετρήσουν ως προθεσμία από την έγκριση του νόμου, του κανονισμού και όχι από μια συγκεκριμένη κάποια άλλη ημερομηνία άσχετα από την έγκριση του κανονισμού. Νομίζω απόλυτα νόμιμο και θεμητό αυτό το αίτημα. Από πλευρά συναδέλφου που αναφέρθηκε το γεγονός ότι οι ηλεκτρικές υποδομές αυτές είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα αυτό το σχόλιο επίσης εφαρμόζεται και, σε άλλα, ε, και, και ε, έχει σχέση και με άλλα σχόλια. Οι υποδομές είναι σίγουρα το πιο σημαντικό. Θα έχουμε αύξηση των ενεργειακών αναγκών και οι προβλέψεις είναι ότι και τα τιμολόγια θα αυξάνονται μέχρι το 2030. Μόνο από το 2030 και μετά με ε, ε, την επίπτωση των επενδύσεων κάτι μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε λοιπόν ότι το φυσικό αέριο θα είναι ένας άρρηκτα συνδεδεμένος εταίρος για τα ενεργειακά θέματα. Το λέει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι πραγματογνώμονες απόλυτα συνδεδεμένο με τις ηλεκτρικές υποδομές, το φυσικό αέριο. Είναι το πιο εύκολα διαθέσιμο, το πιο ελαστικό, το πιο ευέλικτο μέσο και σε σχέση με την ανάλυση κόστους ωφέλους πολύ αποτελεσματικό για το μέλλον. Έχουμε φυσικά και προβλήματα εκπομπών ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα, άνθρακα γενικά. Και για την οικολογική χρήση θα πρέπει η σύλληψη, η αποθήκευση του άνθρακα που βρίσκεται στα σπάργανα ακόμα, στα πρώτα βήματα, θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Και αυτό σημειώνουμε όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πολλά αναμένονται ακόμα σε σχέση με τις εξελίξεις αλλά και για τις χώρες που έχουν πριτανεύοντα ρόλο όσον αφορά κύριο ρόλο του άνθρακα ή του λιθάνθρακα ενεργειακά πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Τώρα, ο συνάδελφος Σόσα Βάγνερ θεωρεί από πλευράς του ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει συνένεση γενικότερη. Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Να υπάρξει συνένεση που είναι θεμελιώδους σημασία. Και γι' αυτό εμείς ε, το αναφέρουμε αυτό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ευθύ εξ αρχής. Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στο θέμα της αποθήκευσης, αποθήκευση ε, νερού. Τελευταίο σημείο. Έχουμε μια τροπολογία σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρούσε ότι η αποθήκευση νερού δεν θα έπρεπε να αναφέρεται στα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος ή συμφέροντος. Και εμείς θεωρούμε πως όχι. Όμως η αποθήκευση αυτή έχει χρήση και είναι ωφέλιμη για τον παραγωγό ηλεκτρικής ε, ενέργειας. Υπάρχει όμως μια αποθήκευση και εδώ υπάρχει ε, το θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την, ε, τα θέματα παραγωγής. Λοιπόν, αυτό να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ λοιπόν τελικά για τις παρεμβάσεις όλων και έχουμε πολλή δουλειά να αναπτύξουμε ακόμα. Ευχαριστώ για την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το fair play, τον, το δίκαιο τρόπο με τον οποίο δέχονται τις τροπολογίες μας, κάποιες από τις τροπολογίες. Ελπίζω θα πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό εύχομαι. Ευχαριστώ. Bene. Ωραία. Πέμπτη 26 Απριλίου στις 6 για τις τροπολογίες. Και θα συζητήσουμε στις 31 Μαΐου στην Επιτροπή. Ψηφίζουμε. Έχουμε καθυστερήσει. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε στα χέρια σας την κάρτα ψηφοφορίας. Ας κάνουμε ένα τεστ. Λοιπόν, μια δοκιμή. Ρούμπιχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να αναφέρω το ότι κανονικά τις ψηφοφορίες μας τις κάνουμε στη δεύτερη ημέρα της συνάντησής μας ε, στην ε, Επιτροπή μας και το πρωί γίνονται αυτές τις δεύτερη ημέρες. Θα διατηρήσουμε αυτή την παράδοση. Τι γίνεται. E Έτσι ήθιστε και θα συνεχίσουμε. δεν είχαμε για σήμερα το πρωί ήταν απλώς ότι δεν είχαμε, βρήκαμε άλλη ημερομηνία που να συμπίπτει με τις δυνατότητες της Επιτροπής Μεταφορών. Πάντως ο κανόνας μας είναι αυτός. Λοιπόν είμαστε εντάξει με την ε, δοκιμή. Οι αριθμοί είναι εντάξει. Ωραία. Αρχίζουμε. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη λέει η Πρόεδρος Έκθεση Νίμπλερ για το roaming. Συμβιβαστική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές νομοθε... εγκρίνεται ομόφωνα ηλεκτρονικά το νομοθετική πράξη Δύο ΕΛΚ παραπάνω. Ωραία, δεν ψηφίζω εγώ. Εγκρίνεται 54 υπέρ και μία αποχή. Δεν είναι εδώ. Συγχαρητήρια κυρία Νίμπλερ.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ με προφορική τροπολογία. Συγγνώμη.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 Un πεπέ di troppo ancora. Ένας ΠΠΕ παραπάνω, ένας ΕΛΚ παραπάνω. Ένας. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. 54 υπέρ, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Bene, passiamo alla relazione della collega Maria Badia Couchet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 Πέρας ψηφοφορίας. Όλοι υπέρ. Κόσμε, κόσμε, κόσμε. Τροπολογία 12. 12. Οχτώ το πρώτο τμήμα λέει τώρα η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28. Έλεγχο πού? Στη 17. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. 47 υπέρ 5 κατά 2 αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα σε μια άλλη γνωμοδότηση της κυρίας Μαρία Μπαντία. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 για μένα απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. 14.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 37 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην 23. Ε, πέρα στις ψηφοφορίες. εγκρίνεται. Η 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 27 30 υπέρ 26 κατά. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα Τροπολογία 10. Πέρα στις ψηφοφορίες. 32 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ Έντεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 54 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τελευταία ψηφοφορία. Έκθεση Κόβατς. Μια ενιαία ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 53 υπέρ, ένας, ε, μία αποχή. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα. Ευχα... Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Συγγνώμη για καναλαθάκι, αλλά πάντα εμείς κοιτάμε αριστερά-δεξιά και υπολογίζουμε. Τι έχουμε τώρα. Allora, passiamo al punto numero 20. 20. Να περιμένουμε λίγο. Δύο λεπτά. Always miss one.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 Bene, mi sembra che sia tornato il silenzio e quindi possiamo continuare. Επανήλθε η ησυχία. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Είμαστε στο σημείο 20 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι με την έκθεση που έχουμε στα χέρια μας πάμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά διότι απλά και τώρα στην κρίση χρέους αυτό που θέλουμε είναι να καλυφθούν αυτά τα ποσά, να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα χρήματα και πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργηθούν νέες καλοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης και γι' αυτό χρειαζόμαστε ικανούς, καλά καταρτισμένους και εκπαιδευμένους επιχειρηματίες, κυρίως επιχειρηματίες γυναίκες. Και διαπιστώσαμε ότι οι νέες αυτές επιχειρήσεις είναι εκείνες που πιο γοργά προσλαμβάνουν στελέχη και προσωπικό. Και εδώ πρέπει να δούμε τις προοπτικές για τη διασφάλιση του μέλλοντος για τις θέσεις απασχόλησης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε πάει με την Επιτροπή Ήτρε στη Βραζιλία και είχαμε και ένα γύρο εκπροσώπων επιχειρήσεων που τους ρωτήσαμε τι θα κάνατε εσείς ώστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εξαγωγή και στην βιομηχανία να ενισχυθούν στην ανταγωνιστικότητά τους και να ανακουφιστούν από γραφειοκρατικά βάρη. Το πρώτο που θα ευχόντουσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περισσότερες πληροφορίες για δημόσιες προμήθειες, δημόσιες συμβάσεις, για τις ανάγκες που υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν. Πληροφορίες και ανακοινώσεις όταν έχουμε νέες υποδομές, για παράδειγμα χρειάζονται νέες επενδύσεις και ενδιαφέρονται για τα clusters, ε, να γνωρίζουν τι συμβαίνει σχετικά. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να περάσουν και να πολιθούν αυτά όσον αφορά και τις δράσεις αυτές και τα προϊόντα. Το δεύτερον, προγράμματα ανταλλαγής. Τους εξήγησα ότι η Επιτροπή Ήτρε ανέλαβε πρωτοβουλία για το πρόγραμμα Έρασμος για νέους επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες. Να προαχθεί λοιπόν αυτή η ανταλλαγή σε μεγάλο πλαίσιο, ώστε να ασχοληθούμε πολύ πιο έντονα ώστε οι νέοι, νέοι άνθρωποι από την Ευρώπη να περάσουν σε αυτές τις χώρες, ώστε επιτόπου να δημιουργήσουν δίκτυα και αυτές οι γνώσεις να περάσουν και στις χώρες τους και να βρουν απήχηση. Και από την άλλη πλευρά, σε αυτές τις τρίτες χώρες, από αυτές τις χώρες φοιτητέ και επιχειρηματίες να έρθουν σε εμά στην Ευρώπη για να τους δείξουμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν εδώ για αυτούς. Για όλα αυτά χρειαζόμαστε την αναγνώριση των διπλωμάτων και πτυχίων σπουδών, την διεθνή αναγνώριση και ισοτιμία τέτοιων πτυχίων και διπλωμάτων. Αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την blue card, για την κιανή Black κάρτα. Εδώ υπάρχει ένας τομέας στις διμερείς συμφωνίες να μεριμνήσουμε οπωσδήποτε ώστε να προχωρήσει αυτό το σκέλος, να προαχθεί ιδιαίτερα. Τρίτο ή τέταρτο, χρειάζονται από πλευράς τεχνικής, τεχνολογίας, στην κατάρτιση, εκπαίδευση κατάρτιση, στην υλοποίηση όλες οι προσπάθειες να ενισχυθούν σχετικά, ώστε να υπάρξει αναγνώριση πιστοποιητικών που θα δίνουν τη δυνατότητα σε θεωρήσεις διαβατηρίων να βρίσκει αυτό την απήχησή του και να αποσαφινιστούν όλες οι συναφείς παράμετροι. Εδώ είναι μια κέρια πρόκληση αυτή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να καλύψουμε. Πρέπει εδώ να μεριμνήσουμε και να δούμε πώς διεθνείς επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν ε, α, τα στελέχη και τις, ε, τους όσους τους τροφοδοτούν ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Και τέλος για τους Ευρωπαίους που εργάστηκαν στη Βραζιλία να ασχοληθούμε περισσότερο με θέματα φορολογικά, φορολόγησης η αρνητική αντιμετώπιση σε σχέση με διπλή φορολόγηση, συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο. Ενδιαφέρονται να δουν και να μάθουν τι γίνεται από πλευράς των ευρωπαϊκών αρχών και DG Tax. Τι μπορεί να γίνει ώστε με την DG Trade, τη Γενική Διεύθυνση για τα θέματα εμπορίου, να δουν τι μπορεί να γίνει ώστε να μην έχουν αρνητική διακριτική μεταχείριση φορολογικά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οικονομικά να τύχουν υποστήριξης από εμάς, ιδιαίτερα με εγγυήσει ε, με εγγυήσει όσον αφορά πιστώσεις και δάνεια. Είναι σημαντικό να μεριμνήσουμε για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν πρόκειται για κεφάλαιο κινδύνου η αξιοπιστία αυτών των ε, επιχειρήσεων πιστοληπτικά να ενισχυθεί, να τονωθεί. Όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών ή για τα κράτη-μέλη μόνο, αλλά ιδιαίτερα για θέματα διαμεθοριακών, διασυνοριακών ε, επαφών και εξαγωγών και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό ώστε να υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση σε αυτές τις ανάγκες, για αυτές τις Πρέπει να είναι προτεραιότητα, ιδιαίτερη προτεραιότητα για μας. Τέλος, τέλος, το αποτέλεσμα μόχλευσης, ποιο θα είναι αυτό που θα πετύχουμε με αυτά τα μέσα ή μέτρα. Πρέπει εδώ να υποβληθούν προτάσεις από πλευράς μας. <clears throat> Για τις παραδοσιακές τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερα θελκτικό να, ε, έχουμε, να υπάρξουν τέτοια θέματα εγγυήσεων ε, ε, ή διασφαλίσεων, διότι πρώτα θέλουν να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα και μετά να δουν ποια είναι τα προτερήματα σε σχέση με επιχειρήσεις που θα εξαρτηθούν από αυτές. Τώρα είναι όμως η θετική χρονική στιγμή, ώστε μέχρι το 2020 σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο να, δούμε, να ξαναδούμε τα κέντρα βάρους που θα θέσουμε και η Επιτροπή Ήτρα διαδραματίζει φυσικά ένα σημαντικό ρόλο για το μέλλον της Ευρώπης ως αυτά. Ευχαριστούμε η κυρία Γιόνισον. Ευχαριστώ λέει ένας κύριος, ευχαριστώ τον κύριο Ρούμπικ για την προσέγγιση του. και τη συνεργασία μεταξύ των σκιωδών. Όλοι νομίζω συμφωνούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχείρηση είναι κάτι το ζωτικό για την οικονομία μας και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε περισσότερα, ιδιαίτερα σε αυτή τη σύγχρονη, την τωρινή ατμόσφαιρα της κρίσης. Η έκθεση αυτή καθώς και η επόμενη του κυρίου Γκρόιτσμαν θα συμβάλλουν νομίζω θετικά στη συζήτηση. Χαιρετίζω το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ρούμπικα, αλλά έχω και μερικά σχόλια που θέλει να κάνει η ομάδα μου και να καταθέσει μερικές τροπολογίες για να βελτιώσει το κείμενο. Θα σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες μας για την υποστήριξη των υπηρεσιών Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν πρέπει πριν τα τέλη του 2012 να αρχίσει να εφαρμόζεται η, ιστοσελίδα, η πολύγλωση στο σελίδα και για την παιδεία θέλω να τονίσω τη σημασία της προώθησης του προγράμματος Έρασμος για τους νέους και για τους νέους επιχειρηματίες για την πρόσβαση στις αγορές συμφωνούμε ότι χρειάζεται περισσότερη στήριξη για να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών ιδιαίτερα μέσω μιας, ενός βελτιωμένου επιχειρηματικού δικτύου στην Ένωση. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι επίσης μεγάλος φραγμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί οι τράπεζες διστάζουν να δανείζουν χρήματα και χρειαζόμαστε και άλλα πρότυπα και παραδείγματα, υποδείγματα χρηματοδότησης. Να συνδέσουμε ας πούμε τις δραστηριότητές τους με το Horizon και άλλους τέτοιους τρόπους. Η γραφειοκρατία πρέπει να μειωθεί και η νομοθεσία να βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως προβλέπει παραδείγματο χάρη η τελευταία οδηγία για τις πληρωμές που δεν έχει ακόμη αρχίσει να εφαρμόζεται. Είναι καλή αρχή αυτή η έκθεση και γι' αυτό θα τη δεχτούμε με μερικές τροπολογίες και προσβλέπουμε σε περισσότερη συνεργασία με τους συνεισηγητές. και να είμαστε όλοι περήφανοι για το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ακριβώς και ο προλαλής σας, θα ήθελα και εγώ σε σχέση με την ε, πρόταση αυτή να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρούμπικ και να προαναγγείλω ότι και εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε από πλευράς μας όπως μπορούμε. Αλλά υπάρχουν και κοινά στοιχεία και σημεία. Κάποια από αυτά θέλω να τονίσω. Το Enterprise Europe Network δεν είναι μόνο στον τομέα της παγκοσμιοποίησης και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερης σπουδαιότητας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση μόνο τότε μπορεί να προαχθεί, να προχωρήσει επιτυχώς όταν το ΕΕΝ μέσα στα κράτη-μέλη έχει επαρκώς ισχυρή βάση. Και πρέπει εδώ απλά να διαπιστώσουμε ότι σε κάποιες περιφέρειες το Enterprise Europe Network έχει πολύ καλά αναπτυχθεί και είναι προσπελάσιμο και εύκολα προσβάσιμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε άλλες περιφέρειες υπάρχει μία και μόνο θηρίδα, one stop shop, ώστε θα πρέπει για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην παγκοσμιοποίηση ε, δυσχεραίνεται πολλές φορές ίσως η πρόσβαση. Αυτή την πτυχή θα πρέπει να την εξετάσουμε λοιπόν αυτή τη συνιστόσα. Δεύτερον, κάνετε λόγο συνάδελφε Ρίμπικ για ορθολογική χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού όσον αφορά και το κόσμε για παράδειγμα και τις δυνατότητες. Είχε εξεταστεί δυνατότητα και σήμερα το πρωί να, υπάρξουν, να υπάρξουν κάποιες διαγραφές. Εμείς νομίζω δεν πρέπει να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Πρέπει να δώσουμε μάχη αυτά τα κονδύλια να αυξηθούν ακόμα και όχι να μειωθούν ή να διαγραφούν. Τρίτον, αναφέρεται στο σημείο 14 της προτάσεις της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύστημα τυποποίησης. Απλά και μόνο θα ήθελα να παρατηρήσω και να πω ότι πιστεύω σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε πιο ξεκάθαρη γλώσσα να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά την εκπροσώπηση συμφερόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του συστήματος τυποποίησης. Είμαι απόλυτα σύμφωνος και θέλω να το αναφέρω ρητά αυτό με το θέμα του ισχυρού κέντρου βάρους που τίθεται στον ορισμό των SME και να μην υπάρξει αποδυνάμωση του ορισμού αυτού με την εισαγωγή για παράδειγμα μιας νέας κατηγορίας. Επίσης συμφωνώ με τις σαφείς ενδείξεις και τοποθετήσεις σας για το ότι όσον αφορά τις μικροεπιχειρήσεις ο αποκλεισμός τους από τις ε, διαδικασίες δεν είναι η πιο συνετή προσέγγιση θα χαιρόμουν αν θα μπορούσαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή να συμφωνήσουμε σε αυτές τις προτάσεις ε, που υποβάλλουμε. Τελευταίο, εκεί όπου το εδάφιο 27 γίνεται λόγος, κάνετε λόγο για ανταγωνιστικότητα, competitiveness, πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν να βρούμε την σύνδεση μεταξύ ανταγωνισμού, καινοτομία, innovation και sustainability και φορείας. Και τέλος έχω και κάποιο πρόβλημα με το εδάφιο 31 από πλευρά σας. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος αν πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει οδικό χάρτη ε, roadmap για αυτό το θέμα και όσον αφορά και την φορολόγηση. Δεν είμαι βέβαιος αν χρειάζεται καν ε, οδικός χάρτης για ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορολόγησή τους. Πρώτον, για το ότι έχουμε εδώ θέματα άλλα από τη φορολόγηση. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη στην χρησιμοποίηση, στην χρήση των βέλτιστη χρήση των κονδυλίων δεν θα είχαν ακριβώς αυτό το συμφέρον. Και αν ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση τότε αυτά που ο Επίτροπος Ποτόσνικ και το Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων έχουν προτείνει, δηλαδή να δούμε την διασύνδεση μεταξύ της ελάφρυνσης της άμεσης φορολόγησης και μιας μετάθεσης του φορολογικού βάρους στην φορολόγηση των ε, περασμένων ε, φορέων και υλικών ε, ενεργειακών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφο Στόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόνο λίγες παρατηρήσεις. Έχουμε συναδέλφους ε, του Ρούμπιχ, τον Ρούμπιχ, ε, την Έρτζοκ που είναι μέλη σε, ενός intergroup για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και συζήτησαν και με τους άμεσα ενδιαφερόμενους τις μυθικές πια ΜΜΕ έχουν άμεση επαφή με τους ε, χρήστες παρατηρήσεις και συγχαρητήρια. Πιστεύω η πρόταση του κυρίου Ρούμπιχ ε, ε, καλύπτει πολλές πλευρές, είναι ιδιαίτερα ανοιχτή η σύμφωνη να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, την πρόσβαση στην αγορά των ΜΜΕ. Για να κάνουμε όμως κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να έχουμε μία μεμονωμένη προσέγγιση. Χρειάζεται μία ευρύτερη προσέγγιση. Όμως ε, θα πρέπει η πρότασή μας ε, όσο ευρία και να είναι να έχει αναφορές συγκεκριμένες σε προγράμματα, σε σχέδια για να μην είναι μόνο ευχές και γενικές ιδέες όλα όσα θα προτείνουμε. Πρώτα απ' όλα να σταθώ στο θέμα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις να μεγαλώσουν, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά τους των ΜΜΕ, αγκυροβολημένες στην ε, επικράτειά τους, να τις βοηθήσουμε λοιπόν για την ανάπτυξή τους, για το μεγάλωμά τους ε, καινοτομία. Χρειάζεται τεχνολογική, διαχειριστική καινοτομία και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία στοχεύουν στη βοήθεια των ΜΜΕ, να βοηθήσουμε για τις νέες αγορές, για, τις, για το διοικητικό κόστος και τη μείωσή του, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε πολλές χώρες και στη δικιά μου το ενεργειακό κόστος βαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους. Το θέμα των πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε τη σχετική έκθεση για την πληρωμή των χρεών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την προθεσμία, αλλά αυτό δεν τηρείται πολύ και ο Επίτροπος Ταγιάννη θέλει να επιμείνει σε αυτό. Μετά έχουμε και την την, το κόσμο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα θέματα ε, του χρέους η υποστήριξη, δεν, για να σταθώ σε αυτό που είπε και ο κύριος Μπουτικόφερ, δεν λειτουργεί πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο. Πολλές φορές έρχεται μία πληροφορία στις Βρυξέλλες, αλλά δεν γίνεται τακτικά. Πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν μία αναθεώρηση. Πριν από μερικά χρόνια το είχαμε ζητήσει, όταν δεν υπήρχε το δίκτυο, αλλά είχαμε άλλα γραφεία που δεν θυμάμαι πώς λεγόντουσαν. Είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να μας κάνει μία έκθεση. Άλλοι είχαν τα εμπορικά επιμελητήρια, άλλοι είχαν άλλους οργανισμούς, άλλους τους πληρώνανε η Ευρώπη, άλλους ε, άλλοι. Και υπήρχε μία τεράστια σύγχυση και δεν ξέραμε τι κάνει, τι, ποιος κάνει τι. Και είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρχει μία σαφή Πίνια, δεν, όχι ένα καπέλωμα, αλλά τουλάχιστον ε, ίδιες προδιαγραφές ε, για τα σημεία αναφοράς. Γιατί πολλές ε, φορές τα προγράμματά μας σταματούν στα δίκτυα επαφής. Εμείς είμαστε έτοιμοι πάντως να σας υποστηρίξουμε. κυρία Φόρντο. Ευχαριστώ. Ξεκινώ ευχαριστώντας τον εισηγητή για την εξαιρετική εκκίνηση. Ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οικονομίες μας. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για το πνεύμα του επιχειρήν από την Ευρωβουλή και για τα ωφέλη όσον αφορά την φορολόγηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρότι η φορολόγηση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να το, να το ξέρουμε αυτό. Χαίρομαι για το ότι θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετώπιση γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων, μείωση του γραφειοκρατικού προσκόμματος και, δυσκολίας, και δυσκολιών δεν θα είναι όλε οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις αυτές που θα εξάγουν. Πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνες όμως που θα δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει να δούμε ότι δεν θα επιληθούν όλες οι ανάγκες όλων ταυτόχρονα. Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε όλες τις ανάγκες και πτυχέ των πολυμορφοποιημένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα, πρέπει να υπάρξει ένα πολύ πιο ζωγόνο στοιχείο σε σχέση με το μέλλον χρειάζεται να ενταχθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών των κρατών μελών η προσπάθεια αυτή. Χαίρομαι για το ότι το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να θεωρείται σαν ένα πιο σημαντικό ε, τμήμα ε, της ζωής μας Προσωπικά θα έλεγα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που θα μπορούσαν να εξαιρούνται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εκτός αν πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν. Τώρα, για τις μεγαλύτερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το κόστος ε, λειτουργίας τους Ίσως αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα. Για τις πραγματικά πολύ μικρές επιχειρήσεις πρέπει να είμαστε ε, ευέλικτοι ώστε να χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτά τα οποία πρέπει να εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο. Η προσπελασιμότητα έχει σημασία σπουδαία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τα δάνεια, πιστώσεις κτλ μπορεί να υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα σε σχέση με τη δημόσια χρηματοδότηση, να δούμε κάποιες εφάντασες δημιουργικές λύσεις που μπορούν να ακολουθηθούν. Angel, χρηματοδότηση Angel, peer financing, supply credits, πιστώσεις εξοπλισμού να δούμε ιδιαίτερα και τον ε, σκιώδη τομέα τον τραπεζικό. Δεν είναι όλες οι δραστηριότητες αυτές υποχρεωτικά αρνητικές, υπονομευτικές. Πρέπει να είμαστε υπέρ των ευφυών δημιουργικών λύσεων για τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. Μου αρέσει η ιδέα σας για το έπαθλο όσον αφορά την καλύτερη εφαρμογή από τους πρώτους, από τις πρώτες. Αλλά το να τιμούμε κάποιους πρέπει να μας κάνει να δούμε και την ανάγκη να κατονομάζουμε και άλλους που δεν θα είναι τόσο, ε, δεν θα συμμορφώνονται να δείχνουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα, διότι το κόστος στους καταναλωτές, τα βάρη στις επιχειρήσεις μας κάνουν να χωλένουμε στην ανταγωνιστικότητα και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και εμείς ως Επιτροπή πρέπει να το σταματήσουμε. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με τους συγητές οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Δύο λεπτά ο καθένας, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυρία Μπούλφκοκ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή υποβάλλεται η πρόταση να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις ε, όσον αφορά τους όρους απασχόλησης, για παράδειγμα στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό σίγουρα είναι μια βελτίωση σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, από την άλλη πλευρά είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι με αυτή την πρόταση ανοίγουν πόρτες και παραθύρια για αρνητικότερες ε, συνθήκες εργασίας ε, για τους εργαζόμενους. Η προστασία πρέπει να ισχύει όμως για όλους τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Θέλουν όμως να υπάρξει απλούστευση και απελευθέρωση λέει της νομοθεσίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι υπό χειρότερους όρους και προϋποθέσεις θα προσλαμβάνονται και θα εργάζονται οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και εμπορικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και ο εισηγητής μας ανέφερε ποια είναι τα προβλήματα των ΜΜΕ που αποτελούν το βασικό κορμό του εμπορίου και είναι και το 85% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2002 μέχρι το 2010 αποτελούν πηγή απασχόλησης Πρέπει να τις βοηθήσουμε να έχουν μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική μέσα στη στρατηγική 2020 με βασικούς στόχους και προτεραιότητες. Θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και στις εθνικές αγορές και στην αγορά της Ένωσης, να έχουν ευκαιρίες στην αγορά στη διερεύνηση των αγορών, να μειώσουμε το διοικητικό άχθος, να βοηθήσουμε το διάλογο, να αναλύσουμε και να καταστήσουμε έχουμε μια σαφή εικόνα και τις τυπολογίες των υπαρχουσών ΜΜΕ. Η Κομισιόν μας παρουσιάζει πολύπλοκα μέτρα και μπορεί να μην είναι και τόσο αποτελεσματικά. Να ρωτήσω λοιπόν την Κομισιόν πρώτο, ποιες είναι οι βελτιώσεις ή υποστήριξη των ΜΜΕ για την πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών, όπως έλεγε ο εισηγητής, και για να, τι κάνουμε για να βελτιώσουμε τον συντονισμό των διαφόρων πρωτοβουλειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα θέλω να ακούσω η Κομισιόν τι λέει. Ευχαριστώ η κυρία Χέρτζοκ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ότι από τους σοσιαλιστές η σκιώδης αρμο... Ε, εισήγηση ε, έχει δοθεί σε εμά και χαίρομαι ότι ε, από πλευρά του κυρίου Ρούμπιχ και για τις προτάσεις που αναφέρονται. Κάποια πράγματα θέλω να αναφέρω. Το πιο σημαντικό πρώτο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην μεταθέσουμε τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το επίπεδο των κρατών μελών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τα του οίκου τους, τα καθήκοντά τους είναι υπόθεση των κρατών μελών κυρίως τι γίνεται με τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά είναι συμπληρωματική, παραπληρωματική τα κράτη-μέλη να μην θεωρήσουν ότι δεν χρειάζεται η δράση τους γιατί τώρα θα τα κάνει όλα η Ευρώπη με τα ε, περιορισμένα κονδύλια που υπάρχουν. Λάθος αυτό. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τα πάντα. Ακόμα και αν δαπανούσαμε όλο τον ευρωπαϊκό προπολογισμό στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, πρέπει να δούμε την αναλογία των αριθμητικών μεγεθών. Θα μπορούσαμε να έχουμε χ μικρομεσαίες επιχειρήσει, μεγάλο αριθμό σε σχέση με το παρελθόν. Αν συγκρίνουμε όμως αυτόν τον αριθμό συνολικά με όλε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεράστιο το βάρο και δεν είναι δυνατόν εμεί να το επομισθούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να απεμπολίσουν αυτή την ευθύνη τα κράτη-μέλη. Καλούμε λοιπόν, πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν σωστά, να αναλάβουν τα των ευθυνών τους. Ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος και για προγράμματα συγχρηματοδότησης. Είναι σημαντικό όταν δίνουμε υποστήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα ε, για το επιχειρήν να ε, συνεισφέρουμε εμείς αλλά να συνεισφέρουν και τα κράτη-μέλη, να μην το αγνοούν αυτό συμφωνώ με αυτούς που ανέφεραν τις δοκιμασίες ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων SME test πολύ σημαντικό αυτό αλλά το τι δαπανούμε και πώς το δαπανούμε είναι σημαντικό να το εξετάσουμε είναι σημαντικό να διατυπώνουμε αυτό το ερώτημα θα ήθελα να πω δύο λόγια για κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Συμφωνώ με τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται βέβαια στην έκθεση, αλλά υπάρχουν κάποιοι τομεί όπου έχουμε πολύ περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει στον τομέα των οικοδομών. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να παγκοσμιοποιηθεί αυτός ο τομέας, άλλες ε, δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα για παράδειγμα, για τον τομέα τον οικοδομικό. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που θα ήθελα να αναφέρω. Συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που έγιναν και να συμπεριλάβουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μας να συμμετάσχουμε. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ακούω τόσο πολλούς να συμμετέχουν στη συζήτηση και να συγχαίρονται όλοι τον Παύλο για την καλή του δουλειά. Αυτό ανταποκρίνεται στο ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη μόνο από μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να έρθει. Γι' αυτό λέγονται ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Ευρώπη. Τώρα, Μια κατηγορία που έχει τόσο μεγάλη σημασία δεν είναι απλώς κατηγορία, είναι σχεδόν το σύνολο της οικονομίας και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει τουλάχιστον οι μικροεπιχειρήσεις λιγότερο από 10-15 υπαλλήλους να, αυτές να έχουν μια χωριστή κατηγορία. Η γραφειοκρατία είναι πρόβλημα βέβαια και οι χρηματικές ενισχύσεις, οι επιχορηγήσεις από την ΕΚΤ πρέπει να δίνονται με αυστηρά ελεγμένα κριτήρια, να δίνονται δηλαδή πράγματι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το αξίζουν και που δεν έχουν νοθευμένο ισολογισμό. Οι επιχειρηματίες συμπεριλαμβάνουν και γυναίκες. Το δείχνουν αυτό πολλές, πολλά στατιστικά στοιχεία και ε, οι γυναίκες επιχειρηματίες ίσως να προωθούν την ανάπτυξη και περισσότερο από τους υπόλοιπους. Θα θέλαμε λοιπόν λίγα περισσότερα και γι' αυτό τέλος. Ως εισηγητής για την ομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχω συζητήσει και εγώ με εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ως προς το θέμα αυτό θα εξισωθούν με τις μεγάλες για να τύχουν τη συμπεριφορά που τους αξίζει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ρούμπιχ για το τόσο ενδιαφέρον έγγραφο. Εγώ θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Λυπούμε που αυτό το οποίο είχαμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τις ευρωπαϊκές ε, πλατφόρμες που θα έπρεπε να δώσουν στα κλάστερ ό,τι τους έλειπε, δηλαδή το να μπορέσουν να κάνουν οικονομή, ε, καινοτομία για τους ίδιους και να βοηθήσουν τις, ε, πιο, τις ε, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν ως υπεργολάβοι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων να ανεξαρτητοποιηθούν και να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κι αλλού, σε άλλες βιομηχανίες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό, όχι μόνο όταν μιλάμε για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά όταν μιλάμε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι εδώ πρόκειται για την δυνατότητα του να κάνουν, να κάνουν καινοτομία κατηδίαν και να μπορούν να βοηθούν και στις επαφές τους με τα πανεπιστήμια, με τα ερευνητικά κέντρα, δηλαδή να έχουν αυτήν την τεχνολογική αυτονομία για να ενισχύσουν αφενός την παραγωγή τους, αλλά απ' την άλλη και όλο το σύστημα, το επιχειρησιακό σύστημα της ε, επικράτειας, το packaging της ε, Μπολόνια, όπου πολλές μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν, παίζουν ηγετικό ρόλο ε, υφίστανται με χιλιάδες όμως από πίσω μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν ως υπεργολάβοι. Ο κύριος Κουκόβιτς, κυρία Κουκόβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρούμπιχ πρώτα απ' όλα. Και αυτό επειδή η αλήθεια είναι ότι αφοσιώθηκε στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι δεν είναι και επίσης θα ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι κακό της ίδιας της πείρας μου. Πρώτα απ' όλα, εκ των ένδων είναι αλήθεια ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις μας και για να γίνει αυτό αν το θέλουμε υπάρχουν πολλά εμπόδια και προσκόμματα στην ενιαία αγορά πρέπει αυτά να άρουμε και να καταργήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα πιο γοργά δεύτερον αν θέλουμε να βασιστούμε, να βασιζόμαστε στο ότι θα υπάρχουν περισσότερες παγκοσμιοποιημένες επιχειρήσεις πάνω από το 13% όπως υπάρχει σήμερα και να διεισδύσουμε στις αγορές της Κίνας, Βραζιλίας και Ινδίας χρειαζόμαστε βελτιώσεις βελτιώσεις στον τομέα των, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Διότι πολλές φορές αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν επωφελούνται από ε, τις πληροφορίες επειδή δεν υπάρχουν διάβλοι και μέσα να, να διαχέονται αυτές τις πληροφορίες. Πρέπει να δούμε ποια κατόφλια πρέπει να ε, μπορέσουν να υπερβούν για να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις. Αν πρέπει να μειωθούν αυτά τα κατόφλια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν με καλύτερες προϋποθέσεις, ας γίνει αυτό. Διότι τις πιο πολλές φορές είναι υπερβολικά υψηλά αυτά τα κατόφλια και παρεμποδίζουν. Πρέπει να λάβουμε επίση υπόψη τα συστήματα εκπαίδευση, παιδεία και κατάρτιση. Σε αυτά πρέπει να εμείνουμε και να επιμείνουμε στο θάρρο, στο ε, ε, στη γενναιότητα, την τόλμη και το επιχειρηματικό πνεύμα. Πρέπει να μπορέσει κανείς να ε, τολμήσει, να έχει γενναιότητα για να μπορέσει να δράσει σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να πείσουμε τις νέους μας ως προς αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε. Η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα διεξήγαγε μια εκστρατεία Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγκρίναμε ένα μανιφέστο. Τρία πράγματα διαπιστώσαμε, συνάδελφε Ρούιμπιχ. Πρόσβαση στις αγορές, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του γραφειοκρατικού βάρους και εμποδίων. Σίγουρα θα σκεφτούμε με, την, με τις τροπολογίες που μπορούμε να καταθέσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να σας υποστηρίξουμε στο εγχείρημά σας σε σχέση με αυτό το θέμα. Δεύτερο σημείο, στη Γερμανία, αλλά και συνάδελφε Ρούμπιχ, νομίζω και στην Αυστρία, έχουμε μια ισχυρή κουλτούρα της α, ανεξαρτησίας και αυτοδύναμης δράσης. Και έτσι λοιπόν έτσι πρέπει να εντάξουμε στον προβληματισμό, προβληματισμό μας και αυτή τη συνιστόσα να αυτενεργούμε αυτοτελώς και αυτούσια. Για παράδειγμα, συζητάμε αυτές τις μέρες ή το, θα το συζητήσουμε στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή τον κανονισμό για τους οικονομικούς ελεγκτές. Και εκεί ο Επίτροπος πρότεινε ότι κεφαλαιακές εταιρείες θα πρέπει να έχουν μια δυνατότητα κεφαλαιουχικές εταιρείες να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εταιρείες ελέγχων. Αυτό όμως θα ήταν μια παρέμβαση στην αυτονομία αυτών των, αυτών των παραγόντων. Μήπως θα άλλαζε λοιπόν κάτι το οποίο θα ήταν μειονεκτικό, μειονέκτημα. Δεύτερον, χαίρομαι που υπάρχει συνένεση. Είδα ότι κατανέβεται αυτό συνεπέρανα και για τα προγράμματα COSME για παράδειγμα, για το πρόγραμμα COSME πρέπει να διαθέσουμε μεγαλύτερες ε, δυνατότητες. Όμως τώρα δεν είναι το θέμα των κονδυλίων όσον αφορά τα κράτη-μέλη που θα απεμπολίσουν τα κράτη-μέλη τις ευθύνες τους το να κάνουν κάτι σε αυτόν τον τομέα. Αν θέλουμε να γίνει κάτι ευρωπαϊκά πρέπει να υπάρχει και ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία στις δράσεις. Στη συνολική συζήτηση που διεξαγάγαμε είδαμε ότι οι επακόλουθοι προβληματισμοί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μας κάνουν να βάλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο και έτσι θα διατυπώσουμε τροπολογίες σε σχέση με το πρόγραμμα COSME και πολύ γοργά μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται μόνο για καινοτομίε, καινοτόμο δράση και high-tech υψηλής τεχνολογίας δράσης για τους στόχους του ορίζοντα 2020 αλλά για πολύ πρακτικά πράγματα. Αν θα μπορούσαμε τα επακόλουθα προβλήματα να επιλύσουμε θα διατηρούσαμε πολλές θέσεις απασχόλησης, θα δίναμε νέο αίμα, ζωογόνες δράσεις και θα υποστηρίζαμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ζητώ κάτι να κάνουμε παραπάνω συνάδελφοι για αυτά τα θέματα. Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Και εξίσου σημαντικό είναι να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι τυπικά και μόνο να πει να έχουμε τέτοια τεστ, τέτοιες δοκιμασίες για τις ΜΜΕ, αλλά να υλοποιούνται αυτά τα, αυτές οι δοκιμασίες. Και αν υπάρχει κάποια αρνητική έκβαση σε τέτοιες δοκιμασίες, ή δεν θα έχουμε μια ε, τέτοια πρόταση ή θα την τροποποιήσουμε. Να συναγάγουμε τις συνέπειες λοιπόν και όχι να πούμε «Α, ήταν αρνητικά τα τεστ, τα, οι δοκιμασίες για τις ΜΜΕ και θα αγνοήσουμε αυτή την έκβαση». Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Yes, thank you, Mrs. Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι Ζουλιάν Κεργέ και είμαι υπεύθυνο στη Γενική Τμήματάρχη στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Θα ήθελα να υποστηρίξω την έκθεση του κυρίου Ρούμπικ που θεωρούμε ότι στηρίζει και εκείνο τη δράση και τις προτάσεις της Κομισιόν για, την για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπροστά στην παγκοσμιοποίηση. Σημεριζόμαστε αυτά που ακούστηκαν εδώ το απόγευμα από πολλούς συναδέλφους σας ιδιαίτερα την προτεραιότητα που δίνουν όλοι για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε αγορές και τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Θα θέλαμε επίσης να απαντήσουμε σε μερικά σχόλια που ακούστηκαν και να κάνουμε μερικές αποσαφηνήσεις. Πρώτον, ο κύριος Τζόνσον μίλησε για την νέα πολύγλωση πρόσβαση που θέλουμε να έχουμε στο Ιντερνετ. Εμείς έχουμε ήδη αρχίσει την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, αλλά μέχρι το τέλος του 12 υπάρχει ακόμα μόνο η βασική του δομή. Η πλήρης λειτουργία του θα αρχίσει στις αρχές του 13. Μετά είχε υπάρξει ένα ερώτημα για τον καλύτερο τρόπο να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διεθνοποιήσουν τη δραστηριότητά τους. Το πρώτο τέτοιο σχετικό συμβόλαιο θα υπογραφεί σε λίγο και θα βασίζεται σε έναν κατάλογο μέτρων που ήδη υπάρχουν από τα κράτη-μέλη για τη στήριξη της πιο διεθνούς δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα καταρτιστεί ένας πληρέστερος κατάλογος για να δούμε αν υπάρχουν ελλείψεις στην ισχύουσα νομοθεσία. Εδώ στόχος μας είναι να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των υπαρχουσών δομών για να βελτιώσουμε ό,τι έχει ήδη γίνει σε επίπεδο κρατών μελών για να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δίκτυο Enterprise Europe που ήδη υπάρχει σε 54 χώρες, πολύ πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και για να υποφεληθούμε από χρήσιμες πρωτοβουλίες που υπάρχουν όπως ε, η Υπηρεσία Σύνδεσης Ένωσης Κίνας για εμπορικά θέματα κλπ. Ως προς τη δυνατότητα να υπάρξει ένα έρασμος μόντους και για τους νέους επιχειρηματίες που αναφέρεται στην παράγραφο 13 και ανέφερε επίσης ο κύριος Ντόνσον, η δυνατότητα αυτή έχει εξεταστεί ήδη. Υπάρχουν ορισμένα πρακτικά εμπόδια όμως για την εφαρμογή αυτής της πρότασης και το μελλοντικό πρόγραμμα COSME και το τωρινό SIP δεν έχουν καταφέρει να τα ξεπεράσουν. Υπάρχουν προβλήματα προς τον αριθμό των χωρών που ενδιαφέρονται και των οντοτήτων που μπορεί να χρηματοδοτήσει η Ένωση. Είναι και αυτό μια δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες βέβαια με την Ιαπωνία, την Κίνα ή με τη Βραζιλία που συνδιοργανώνονται με επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ή εφαρμογή δραστηριοτήτων πέρα από τις ήδη υπάρχουσες για ανταλλαγές επιχειρηματιών μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών. Άλλο θέμα, η εφαρμογή της δοκιμής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε πολύ με μεγάλη συνέπεια. Γι' αυτό με εκπλήσει η παράγραφος 17, γιατί εμείς νομίζουμε ότι μία περσινή μελέτη, ε, ότι μία περσινή μελέτη έδειξε ότι η δοκιμή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εφαρμόστηκε πολύ συνεπώς από την Κομισιόν και ως αποτέλεσμα κάναμε πλήρη αξιολόγηση και θέλουμε να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα συστηματικά. Ελπίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, επιτρέπουν, δίνουν χώρο για διαφορετικό, για ποικίλο περιεχόμενο και ποιότητα και η περσινή μελέτη του Κοινοβουλίου είχε πολύ πιο θετικά συμπεράσματα από αυτά που ακούσαμε ή αυτό που γράφει η έκθεση αυτή. Ως προς τον αποκλεισμό των μικροεπιχειρήσεων και εδώ πρέπει να γίνουν να δοθούν ορισμένε αποσαφηνήσεις. Τονίζω ότι από το 2012 η πρόθεσή μας είναι στην προετοιμασία όλων των μελλοντικών νομοθετημάτων μας να αποκλείονται οι μικροεπιχειρήσεις από το εύρος της προτινόμενης νομοθεσίας εκτός εάν υπάρχει η δυνατότητα να αποδειχθεί ότι θα ήταν θετικό κάτι τέτοιο. Στην φάση της αξιολόγησης πρέπει να αποδεικνύεται ότι η νομοθεσία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικροεπιχειρήσεις. Και αν δεν υπάρχει τέτοια απόδειξη θα αποκλείονται από αυτή τη νομοθεσία. Εκεί που πρέπει να καλύπτουμε τις μικροεπιχειρήσεις θα γίνεται θα λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για να ξεπεραστούν όλοι η διοικητική, η νομοθετική, η γραφειοκρατική φραγμή μπορεί αυτές να αντιμετωπίσουν. Για το ερώτημα της κυρίας Τόγια για τη διακυβέρνηση του δικτύου Enterprise Europe, η Κομισιόν έχει συναντηθεί με εκπροσώπους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και προετοιμάζουμε σχέδιο πρότασης για τη νέα διάρθρωση της διακυβέρνησης και ιδιαίτερα το δικαίωμα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων αυτών με τους άλλους εταίρους μας. Άλλο σημαντικό σημείο οι πιθανές αλλαγές του ορισμού μικρομεσαία, της μικρομεσαίας επιχείρησης. Currently, uh, carrying out... Αυτή τη στιγμή κάνουμε μία ανεξάρτητη αξιολόγηση του ορισμού στα πλαίσια του κανονικού και τακτικού ελέγχου που κάνουμε δεν έχουμε καμία πρόθεση ή σχέδιο να κάνουμε να δημιουργήσουμε μια χωριστή κατηγορία όπως τα mid caps αλλά ακούμε ότι μερικοί ζητούν λένε ότι το mid caps θα έχει τα ίδια προβλήματα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν έχουμε βρει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχει καμία εμπορική αποτυχία που να δικαιολογεί δημόσια παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθήκων λειτουργίας αυτού του είδους των επιχειρήσεων. Τέλος, πλην κλείσω, θέλω να υπενθυμίσω την επιστολή του Αντιπροέδρου Ταγιάννη που απαντούσε σε αυτά που ζήτησε ο κύριος Πρόντι γιατί και εμείς συμφωνούμε για τη σημασία των clusters. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρούμπιχ. Μάλιστα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις πολυάριθμες προτάσεις και ιδέες και χαίρομαι για τις τροπολογίες που θα καταθέσετε που και διαπιστώνω ότι λόγω έλλειψης χώρου πολλά δεν μπόρεσα να τα εντάξω στο κείμενό μου που και για μας έχουν μεγάλη σημασία και έτσι θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι προσβλέπω ιδιαίτερα σε αυτές τις τροπολογίες από πλευρά σας για παράδειγμα το θέμα των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τώρα σε σχέση με τα κράτη-μέλη, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και πώς μπορούμε και σε εθνικό επίπεδο να δώσουμε υποστήριξη. Πώς μπορούμε η υποστήριξη αυτή να διαμορφωθεί στο εθνικό επίπεδο, θα πρέπει όλα αυτά να βρίσκονται στο επίκεντρο και είναι 1% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς υποστήριξης. Εδώ αφορά αυτό μια πολύ μικρή ομάδα από τις 25 εκατομμύρια επιχειρήσεις που έχουμε συνολικά ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ευγνώμων θα ήμουν αν θα συζητούσαμε όλα αυτά τα πράγματα σε σχέση με, αυτή τη, με αυτά τα ζητήματα. Τι γίνεται, τι θα γίνεται στις ευρωπαϊκό επίπεδο και σε σχέση και φυσικά και με τις ε, εξαγωγές που διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Τι γίνεται με επιχειρήσεις που δεν είναι ακριβώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορούμε όλα αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσουμε. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικρές τέτοιες επιχειρήσεις που δεν απασχολούν ε, εργαζόμενους. Γιατί δεν απασχολούν εργαζόμενους και συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέφους ότι εδώ πρέπει να υπάρξουν διατάξεις προστασίας των εργαζομένων. Όλα αυτά όμως πρέπει να είναι καλά προσαρμοσμένα σε ένα καθεστώς αμοιβαιότητας. Πώς μπορούμε να πετύχουμε ότι γυναίκες επιχειρηματίες θα προσλαμβάνουν σύμφωνα με όλα αυτά εργαζόμενους. Αν από τις 25 εκατομμύρια επιχειρήσεις κάθε μια προσλάμβανε έναν εργαζόμενο, θα λύναμε το πρόβλημα των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια προβλήματα υπάρχουν και εργάζονται μόνες τους αυτές οι μικρο-μικρο επιχειρήσεις και δεν απασχολούν κανέναν, ενώ είναι ε, αυτοεπιχειρούντες οι ιδιοκτήτες τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά τα θέματα μέσα στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με, νέο, με νέες πρωτοβουλίες. Αυτά πρέπει να δούμε. Χαίρομαι ήδη ε, ε, προσβλέποντας την επόμενη συνάντησή μας. Όλα αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά την έκθεσή μου. Χαίρομαι λοιπόν για τις προτάσεις των συναδέλφων και την επόμενη συνάντησή μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ τον Πόλο Ρούμπιχ. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα. Να θυμίσω ότι στις 8 Μαΐου θα έχουμε μία κρόαση τη Ήτρα για τη ΜΜΕ. 10 Μαΐου για την κατάθεση τροπολογιών το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Τζαβέλα έχει το λόγο. Ε, η διεθνής διάσταση του, της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 υποστηρίζοντας διμερείς και διεθνή, περιφερειακές και διεθνείς εταιρικές σχέσεις στοχεύει μεταξύ άλλων και στη βελτίωση της πρόσβασης της αγοράς ανάπτυξη εμπορικών δυνατοτήτων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αυξημένη ορατότητα της Ένωσης παγκοσμίω. Θα αντικαταστήσει το δημοσιονομικό εργαλείο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και άλλες υψηλών εισοδημάτων χώρες και περιφέρειες. θα έχει πολύ περισσότερο εύρος και γεωγραφικά και θα συμπεριλαμβάνει και τρίτες χώρες. Έτσι θεωρείται σαν ένα στοιχείο στήριξης για την εξωτερική προβολή των ευρωπαϊκών προβλημάτων και ως τέτοια το μελλοντικό αυτό νέο εργαλείο ή υπηρεσία θα συντονίζει πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τον Ορίζοντα 2020 για την έρευνα και την καινοτομία, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας των, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως προέτεινε και η Επιτροπή μας. Τέλος, κάτι διαδικαστικό. Η διορία κατάθεση τροπολογιών παρατάθηκε για να μπορέσουν όλες οι ενδιαφερόμενες επιτροπές να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα. Η εξωτερικών έστειλε επιστολή στη διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών ζητώντας την αρμοδιότητα έναντι της Επιτροπής Εμπορίου και τελικά αποφασίστηκε να δοθεί στην Ήτρα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπαρέα έχει το λόγο, είναι η σκιώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών. Ναι, ναι, είναι πολύ είναι μπερδεμένο το όνομά μου. Τα μέσα για συνεργασία με τρίτες χώρες αποτελούν μέρος της γενικής αρχιτεκτονικής για το εξωτερικό εμπόριο και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, όπως το τόνισε και η συγγήτρια. Ε, άμα συμμετέχει έντονα παγκοσμίω ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βοηθήσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο να προχωρήσει ως προς τις ιδέες και τις αξίες. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο της Κομισιόν που αποτελεί μοχλό για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής πρέπει να εξωθήσουμε την εξωτερική διάσταση, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την έρευνα, την ενεργειακή ασφάλεια, ε, την κλιματική αλλαγή και τα πνευματικά δικαιώματα. Ένα 308 εκατομμύρια λέει η ομιλήτρια. Θα μπορούσαμε με αυτό το ποσό έστω και αν δεν είναι μεγάλο να βοηθήσουμε δίνοντας τη συμπληρωματικότητα στην εξωτερική δράση μέσα από, το πρόγραμμα Κόσμος ή από το, πρόγραμμα, το ερευνητικό πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα. Πρέπει να τονίσουμε την συμπληρωματικότητα με άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Αυτή η έκθεση έχει επιπτώσει σε έναν οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν που θα διατηρήσει ελπίζω το πνεύμα της Λισαβόνας για να μπορεί το Κοινοβούλιο να αποφασίζει ποια θα είναι η συνεργασία με τρίτες χώρες και που μας, πράγμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ την συνάδελφο Μπαρέα. Δεν βλέπω κανέναν άλλο σκιώδη, ίσως εγώ φταίω και δεν βλέπω. Κανένας άλλος δεν ζήτησε το λόγο. Δίνω το λόγο στον κύριο Μέτσες που είναι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ούτε και η Κομισιόν είναι εδώ. Α, εκεί είναι. Θέλει η Κομισιόν το λόγο. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρέμβουμε. Με σύντομο τρόπο για αυτό το θέμα στη μερισία διάταξη δεν θα μακρηγορήσω στα σχόλιά μου. Απλώς να πω ότι η γενική χαρακτήρα αυτού του μέσου όπως προτάθηκε και όπως χαρακτηρίστηκε από τους δύο προλαλήσαντες βρίσκονται όλα πολύ κοντά στις δικές μας αρχικές προθέσεις. Προσεκτικά διαβάσαμε τις τροπολογίες που κατέθηκαν. Θα είναι τώρα συνεισφορά στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν σε σχέση με την Επιτροπή ΑΦΕΤ για αυτό το μέσο. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες στοχεύουν στο θέμα του να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή ατζέντα και τα ενεργειακά θέματα και ο ανταγωνισμός και η καινοτομία όλα αυτά θα αντανακλώνται επαρκώς στο μέσο αυτό και θεωρούμε και εμείς ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το νόημα αυτού του εγχειρήματος, του πρώτου στόχου και στο αντίστοιχο άρθρο γίνεται λόγος για την ενδυνάμωση της διεθνούς συνιστώσας της στρατηγικής του 2020 με στόχο την βελτίωση προσπελασιμότητας στις αγορές, την βελτίωση του εμπορίου, την ενδυνάμωση της Ευρώπης. Και για το θέμα σε σχέση με το μικρό φάσμα κονδυλίων, αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυστηρά να θέσουμε προτεραιότητες στις δράσεις μας για να μπορέσουν με τα με τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα να καλυφθούν. Αυτά τα θέματα θέλουμε να αντανακλώνται και θα πρέπει με το μέσο εταιρικής σχέσης έτσι να δράσουμε. Και θα πρέπει να δούμε, ενώ δεν θα είναι δυνατόν όλα να καλυφθούν σε όλες τις λεπτομέρειες, στα κύρια σημεία τους να δράσουμε έτσι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η συγγήτρια θα ήθελε το λόγο για κάποιο τελικό σχόλιο. Κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω ότι κατατέθηκαν κάποιες τροπολογίες στο παράρτημα αυτό του PI και υπάρχει αναφορά και ε, τονίζεται, τονίζονται οι τομείς της Επιτροπής Ήτρε θα δείτε ότι υπάρχει έμφαση ε, ενδυναμώνονται τα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας και έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες που επικεντρώνονται στα θέματα δικών μας αρμοδιοτήτων μέσα στην Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Αύριο 25 Απριλίου στις 12 η, κατάθεση, η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Επόμενο σημείο, οι βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες ε, που αφορούν στο, πετρέ, σχιστολιθικό αέριο και στο πετρέλαιο. Κυρία Τζαβέλα. Thank you, Madam Chair. Um, shale gas is a είναι θέμα το ΣΕΛΚΑΣ. Πολύ σημαντικό πρόβλημα για την Ευρώπη. Η έκθεση δομείται σε τρία τμήματα. Το ένα είναι το ενεργειακό, το δεύτερο το βιομηχανικό και οικονομικό και το τρίτο τμήμα αφορά τις βέλτιστες πρακτικές και την κοινή γνώμη. Για τα ενεργειακό, την ενεργειακή πτυχή, λέω πόσο σημαντική είναι η Shell Gas για την ενεργειακή μας ασφάλεια. Επίσης, λέμε ότι, στην, ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει και να καταλογογραφήσει όλους αυτούς τους σπόρους που υπάρχουν στην περιφέρειά της. In... Αέριο. Επίσης νομίζω ότι το σχιστολιθικό αέριο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη γενική αγορά του αέριου. Έχουμε πολλά στοιχεία από την παραγωγή σχιστολιθικού αερίου στην Αμερική. Θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη θέση των πελατών εταιριών φωταερίου και μπορεί να οδηγήσει και σε χαμηλότερες τιμές. Η εγχώρια παραγωγή τέτοιου είδους αερίου θα διασφαλίσει περισσότερο την ασφάλεια των προμηθειών γιατί τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα εξαρτώνται από εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες χώρες στις ενεργειακές, για τις ενεργειακές αγορές λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της Ευρώπης και για την οικονομία των κρατών μελών να διασφαλίσουν αν διαθέτουν τέτοιους χιστολιθικούς πόρους. Δεύτερο τμήμα είναι η μετάβαση από την οικονομία χωρίς άνθρακα. Εγώ γράφω ότι αφού η Κομισιόν και όλοι συμφωνούμε συμφωνεί ότι το αέριο θα παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στο ενεργειακό μας σύστημα αφού είναι γρήγορος και φτηνός τρόπος μείωση των πιο μολυντικών ενεργειακών πόρων θεωρούμε και εμείς ότι το σχιστολιθικό αέριο θα μπορούσε σαν μεταβατικό καύσιμο να παίξει ζωτικό ρόλο ιδιαίτερα σε χώρες μέλη που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. Επίσης, αφού μερικές μορφές ανανεωσίμων πηγών ενέργειας όπως ο άνεμος δεν είναι σταθερές και πρέπει να έχουν από πίσω και άλλες πιο βάσιμες πηγές θα μπορούσε το συστολιστικό αέριο να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και ζητούμε από την Κομισιόν σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για την ενέργεια να κάνει αξιολόγηση για αυτού του είδους το νέο τύπο αερίου να το χαρτογραφήσει και τελικά η αγορά να αποφασίσει. Τώρα τα βιομηχανικά και εμπορικά ζητούμε από τη βιομηχανία να προσέξει αυτό το νέο προϊόν στην Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη έχει μεγάλη καθυστέρηση ως προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν έχουμε ειδικευμένου εργάτες και εμπειρογνώμονες για να εκμεταλλευτούμε αυτή την πηγή και γι' αυτό το λόγο σημειώνουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για τον τομέα των υπηρεσιών για να δημιουργηθεί σε αυτό το προϊόν. Έτσι πιστεύουμε ότι οι προσδοκίες για την ταχύτητα ανάπτυξης του σχιστολιθικού αερίου πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Βλέπω ως πρόβλημα την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη για το σχιστολιθικό αέριο. Προτείνω λοιπόν οι χώρες που έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη τέτοιων πόρων στην επικράτειά τους να προβλέψουν και την επιμόρφωση ειδικευμένων εργαζομένων μέσα στο υπάρχον τους σύστημα παιδείας. γιατί και τώρα χρειάζεται να επιμορφώνουν ή να εισάγουν προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες για άλλου είδους εξορίξεις. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να εισαγουν προσωπικο απο τις ηνωμενες για αλλου ειδους εξοριξεις επισης θα ηθελα να τονισω οτι η ενεργειακη πολιτικη πρεπει να αναγνωρισει και να αντιμετωπίσει πιθανούς φραγμούς της επενδύσεις για την ανάπτυξη αυτού του αερίου στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν πράγματι φραγμοί, δηλαδή το πλαίσιο αδειοδοτήσεων. Πρέπει να έχουμε μια προστατευτική αμπρέλα νομοθεσίας ή συστάσεις για τη χορήγηση αδειών για το σχιστολιθικό αέριο που θα μπορούσε να είναι μια νέα μέθοδος αδειοδοτήσεων σε εθνικό επίπεδο. Τονίζουμε ότι σε ορισμένες χώρες μέλη δεν υπάρχει αρκετή διαβούλευση για τις αδειοδοτήσεις και τους ζητούμε να αναθεωρήσουν την νομοθεσία τους και να δουν να φροντίσουν να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης ζητούμε μία μονοαπευθυντική θηρίδα που λένε για να διευκολυνθούν έτσι οι ε, επενδύσεις και τώρα περνάμε στο τρίτο τμήμα. Πρέπει να υπάρξει πλήρης κατανόηση του ενδιαφέροντος που αντιπροσωπεύει για το περιβάλλον το σχιστολιθικό αέριο και καλύτερη κατανόηση και γνώση του τι θα μπορούσε να γίνει για να μειωθούν οι πιθανές αρνητικές του συνέπειες. Η χρήση της καλύτερης τεχνολογίας κτλ. Αλλά κυρίως εποπτεία των εξορίξεων σε όλες τις φάσεις. Επίσης τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι όσοι εξορίσουν να έχουν προηγουμένως πλήρως πληροφορήσει την τοπική κοινότητα περί του πρακτέου, τι χημικές ουσίες θα χρησιμοποιηθούν, δημόσια όλα αυτά, δημόσια, public disclosure που λένε. για τους τρόπους με τους οποίους θα εξοριστεί και επίσης ζητούμε από τις εταιρείες που έχουν αρχίσει τις εξορίξεις να καθαρίσουν τους τόπους των εξορίξεων. Και για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια περί του τι είναι το σχιστολιθικό αέριο, τι σημαίνει και τι επιπτώσεις έχει, προτείνω να διδημοποιηθούν χώρες της Ένωσης με πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν εμπειρία από αυτή την εξόρυξη, πόλεις και χωριά να διδημοποιηθούν για να έχουν περισσότερη και καλύτερη πιο άμεση πληροφόρηση των τοπικών κοινοτήτων. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, η έκθεση μου γράφτηκε στα πλαίσια της Επιτροπής μας και αναφέρεται στο σχιστολιθικό αέριο από την άποψη της ενέργειας και της βιομηχανίας. Τονίζω ποιες είναι οι υποχρεώσεις της βιομηχανίας βέβαια, αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε ακόμα στην Επιτροπή Ήτρε και πρέπει να έχουμε και την ενεργειακή πτυχή. Ευχαριστώ και αν υπάρχουν απορίες να μου τις πείτε. Εγώ τα μελέτησα, τα είδα όλα και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ε, δεν θέλησα να σας διακόψω αλλά μακρηγορήσατε. Εκτιμήσαμε βέβαια την τοποθέτησή σας. Ε, ξεκινάμε με τους Κιώδης. Συνάδελφος Μπρεζίνα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω μεγάλες ευχαριστίες στην εισηγήτρια για αυτή την έκθεση, διότι πιστεύω ότι δεδομένου του συνήθους χώρου ή έκτασης που έχει μια τέτοια έκθεση κάποιων σελίδων όλων και όλων. Η έκταση που αντιμετώπισε το μεγάλο περίπλοκο ζήτημα αυτό και όλα τα συναφή προβλήματα σε σχέση με το σχιστολιθικό αέριο με αποτελεσματικό τρόπο από το δυναμικό που έχει αυτό το προϊόν στις επιπτώσεις στη βιομηχανία και σε όλες τις άλλες πτυχές όπως την πρόσβαση όσον αφορά την, ε, τις βέλτιστες εφαρμογές και πολλά άλλα συναφή θέματα. Και για όλα αυτά σας ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια, κυρία Τζαβέλα. Τούτων λεχθέντων θα ήθελα να πω ότι δεν θέλω να επαναλάβω με κανένα τρόπο όλες τις πτυχές τις οποίες προανέφερε η συγγήτρια. Περιτεύει αυτό σίγουρα. Επιτρέψτε μου μόνο να επαναλάβω ότι κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τους πραγματογνώμονες τα σημεία 7 και 15 αυτής της έκθεσης ήταν εκείνα που αξιολογήσαμε περισσότερο. Εγώ προσωπικά ιδιαίτερα μέσα σε πρακτική και σε επαφές με, το, με την εξόριξη σε μεγάλο βάθος ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τις τροπολογίες της εισηγήτριας. Πιστεύω προσωπικά ότι η καλύτερη τροπολογία, η καλύτερη που ας το πω έτσι αφοπλίζει τα επιχειρήματα πολλών ε, επιφυλάξεων που ακούγονται από περιβαλλοντολόγους είναι η 26α 26α λοιπόν τροπολογία, η οποία αναφέρεται σε τεχνικές δυνατότητες πρόληψης ε, κινδύνων και βλαβών εις βάρος του περιβάλλοντος. Και πιστεύω ότι μια έκθεση με τέτοιο εύρος είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειαζότανε και αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε στην Ήτρε ως σωστή δουλειά. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε το δυναμικό του συστολιθικού αερίου στην Ευρώπη και καλό θα ήταν να μπορούσαμε να υλοποιήσουμε, να, κάνουμε κάποιες, κάποια βασική έρευνα. Όχι μόνο εκτιμήσεις για το δυναμικό και τα αποθέματα αυτού του συστολιθικού αερίου, αλλά να πω και κάτι άλλο. Σε σχέση με τι εφαρμογέ συστολιθικού αερίου, οι τιμέ για παράδειγμα, του φυσικού αερίου ε, σε σχέση με την Ευρώπη που είναι ε, χαμηλότερες αλλού. Εμείς πληρώνουμε στους παρόχους ε, αυτή τη διαφορά. Το όφελος των το συμφέρον των τρίτων χωρών δεν είναι το ότι θα έπρεπε η σχιστολιθική εξόριξη του σχιστολιθικού αερίου να διεξάγεται στην Ευρώπη. Σας το αναφέρω αυτό επειδή είναι μια παρέμβαση. Παρέμβαση στις εμπορικές σχέσεις που υφίστανται στην Ευρώπη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Να το θυμόμαστε λοιπόν αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Κάλφιν για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω και εγώ την κυρία Τζαβέλα για την έκθεσή της. Πράγματι πιστεύω ότι οποιαδήποτε νέα δυνατότητα ενεργειακών πόρων στην Ευρώπη πρέπει να εξεταστεί σοβαρά και αυτή είναι πολύ πολύτιμη πρόταση. Κατανοώ πλήρως τι εννοεί η κυρία Τζαβέλα, δηλαδή ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη βιομηχανική πτυχή, αφού είμαστε η Επιτροπή Βιομηχανίας, αλλά για να γνωρίζουμε πλήρως τα πράγματα πρέπει να γνωρίσουμε ότι σε μερικές χώρες μέλη συζητιέται το πράγμα και υπάρχουν αντιρρήσεις. Πρέπει να το ακούσουμε και αυτό. Αν θέλουμε έκθεση αποτελεσματική πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας γιατί η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει. Πρώτον, να λέγεται κάτι στην έκθεση ρητά ότι το ενεργειακό μείγμα είναι επιλογή της κάθε χώρας. Δεν υποχρεώνεται κανείς να κάνει οποιοδήποτε μείγμα. Δεύτερον, τα περιβαλλοντικά, οι ανησυχίες για το περιβάλλον θα ήθελα να ενδυναμωθούν εδώ και για τις βέλτιστες πρακτικές δεν αρκεί ως παράδειγμα γιατί ε, και εδώ υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις και ε, κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν όλοι μαζί οι υπόψη και να είναι δημόσια. Ορισμένα διαμεριθωριακά προβλήματα υπάρχουν επίσης όταν μιλάμε για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου οι δημόσιες διαβουλεύσεις ε, που γίνονται και πρέπει να γίνουν Ολυμπιακή και είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί και αυτό περαιτέρω στην έκθεση. Πάντως είναι πολύ καλή και βάση για περαιτέρω συζήτηση και ελπίζω να εγκριθεί από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Φιώνα Χολ. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα της Ένωσης να διευθετήσει τα του συστολιθικού αερίου, αλλά και των κρατών μελών. Πράγματι το νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης συζητιέται αν πρέπει να τα καλύπτει όλα ή όχι, αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εχθές η Κομισιόν είπε ότι είναι πρόωρο να καταλήξουμε ότι η ενωσιακή νομοθεσία χορηγεί πλήρη προστασία. Έχουν ευθύνη και οι χώρες μέλη για να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζουν ήδη σωστά και αποτελεσματικά την υπάρχουσα νομοθεσία για το περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να μάθουμε πολλά από τα παραδείγματα που έχουμε για τις υπεράκτιες εξορίξεις πετρελαίου. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, ας πούμε καταλάβαμε από αυτές ότι πρέπει ανατοποθεσία, αναεξόρυξη να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας. Καταλάβαμε τη σημασία που έχει χρήση της καλύτερης δυνατής διαθέσιμης τεχνολογίας αυτό είναι θέμα βελτίστων πρακτικών και κάτι παραπάνω οι ενωσιακές εταιρείες πρέπει να διατηρούν τα πρότυπα που εφαρμόζουν στην Ευρώπη και όταν εργάζονται αλλού. Δεν έχουν όλοι βέβαια τα ίδια πρότυπα, αλλά ελπίζω ότι και για τις εξορίξεις πετρελαίου και για το σχιστολιθικό αέριο θα το δεχτεί αυτό η Κομισιόν. είπε η συγγήτρια ότι είναι μεταβατική, μεταβατικό καύσιμο το σχιστολιστικό αέριο. Πράγματι συχνά λέγεται ότι το αέριο γενικά είναι λιγότερο μολυντικό από τον άνθρακα. Αλλά στην πράξη δεν έχουμε στοιχεία για τις εκπομπές από τα αέρια. Ξέρουμε ότι μπορεί ανάλογα με τη μορφή ενεργείας που χρησιμοποιείται και την τεχνολογίες που χρησιμοποιείται να αυξηθεί η εκπομπή διοξιδίου το carbon footprint. Επίσης υπάρχει το θέμα του πτητικού μεθανίου γιατί μπορεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα μεθανίου να διαφύγει και είναι και αυτό ένας κίνδυνος. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει μελέτη και ανάλυση όλου του κύκλου παραγωγής ή ζωής του σχιστολιθικού αερίου για να είμαστε σίγουροι για τα γεγονότα που θα διαθέτουμε. Τέλος, για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας υπάρχει κάποιο πρόβλημα χρονοδιαγράμματος με το σχιστολιθικό αέριο δεχτήκαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι θέλουμε να κινηθούμε πολύ φιλόδοξα σε μια οικονομία μέχρι το 2015 με όσο δυνατόν λιγότερο άνθρακα. Αλλά ίσως και από το, ε, το 2030, αλλά 50. Ίσως όμως μέχρι το 2030 ήδη να πρέπει να το πετύχουμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα που είναι δύσκολο να δούμε αν και πόσο, κατά πόσον το σχιστολιθικό αέριο μπορεί να αντικαταστήσει άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρισμού μέχρι το 2030. Είναι μια πρόσθετη δυσκολία αυτή. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριος Μπιούτι Κόφερ που είναι ο για τους πράσινους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα πρέπει να πω με την ανάλυση του εισηγήτριας ότι πρέπει να είμαστε άκρος ρεαλιστικοί στις προσδοκίες μας όσον αφορά το σχιστολιθικό αέριο. Όταν αναφέρω αυτό, ιδιαίτερα έχω υπόψη μου τον ρόλο των πολιτών, εκείνων που δεν θέλουν να ισοπεδωθούν από την εξορρυκτική βιομηχανία και τις δραστηριότητές της. Σε κάποιες χώρες ήδη υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με προσπάθειες ισοπαίδωσης, ισοπαίδωμα, ισοπαιδωτικής αντιμετώπισης των πολιτών και στη Γαλλία και στη Βουλγαρία. Με εξέπληξε ότι είπατε ότι ευρέω υποστηρίζετε την έκθεση, διότι πιστεύω ότι πολλοί πολίτες στη χώρα σας είναι πολύ πιο κριτικοί στην τοποθέτησή τους ε, από ότι αυτή η τοποθέτησή σας. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος και αναφέρω δύο θέματα. Πρώτο, το σχέδιο έκθεσης τι λέει. Λέει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρώιμη εκμετάλλευση επαρκεί, είναι επαρκές. Τώρα, αν σωστά θυμάμαι το τι μας είπε η μελέτη που ο Επίτροπος Έτιγκας ζήτησε να συνταχθεί η μελέτη αυτή, αναφέρει και λέει ότι για μια πιο εμβαθυμένη, ευρύτερα ανεπτυγμένη επένδυση στο συστολιθικό αέριο και δραστηριότητες συναφής θα χρειαζόταν, θα έπρεπε να επανεξετάσουμε το σύνολο του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό όμως δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ. Δεν θα έπρεπε ποτέ να λέμε το ίμιση, τη μισή αλήθεια μόνο. Να λέμε την πλήρη αλήθεια, συνολικά. Εξετάζοντας και βλέποντας ότι κράτη-μέλη έχουν συνολικά όλη την ελαστικότητα να το κάνουν αν αυτό προτιμούν, να ακολουθήσουν αυτή την οδό, θα έπρεπε να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στο να πούμε όσο το δυνατόν νωρίτερα θα έπρεπε να βελτιώσουμε αυτό το ευρύ πλαίσιο νομοθετικά, το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεύτερη παρατήρηση. Πιστεύω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να επενδύσουμε και να είμαστε πολύ πιο ξεκάθαροι και αυστηροί στην ορολογία μας για τις χημικές ουσίες και τη διαφάνεια σε σχέση με αυτές και να δώσουμε προτεραιότητα σε τεχνολογίες που αναπτύσσονται και που υπόσχονται την ε, διαρριγμάτωση να την κάνουν, να την επιτυγχάνουν χωρίς χημικές ουσίες. Φυσικά έχουν μελήματα για την υγεία τους οι πολίτες που είναι πάνω-πάνω όσον αφορά τις προτεραιότητες σε σχέση με άλλες επιφυλάξεις τους θέματα υγείας έχουν προτεραιότητα. Αν υπάρχει δυνατότητα διαρριγμάτωσης χωρίς χημικές ουσίες, αυτό νομίζω είναι πολλά υποσχόμενο. Δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι αυτό το καύσιμο, αυτό το ειδικό ξεχωριστό καύσιμο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο προς μια πιο πράσινη μελλοντική προοπτική. Διότι πρέπει να δούμε τον ισολογισμό των ε, αερίων θερμοκηπίου και πρέπει να πω ότι υποστηρίζω αυτά τα οποία ανέφερε η προλαλήσασα να ζητήσουμε να έχουμε μια ανάλυση του συνολικού κύκλου ζωής όσον αφορά τον ισολογισμό το πώς ισοσκελίζεται το θέμα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πιο θετικό όπως αναμένεται ίσως. Και κατά τα άλλα μια συγκεκριμένη πτυχή τώρα, ότι τα πράγματα κινούνται πολύ πίσω από τη ΣΥΠΑ, χωλένουμε πίσω από τη ΣΥΠΑ. Θα έπρεπε να κάνουμε κάθε προσπάθεια να επωφεληθούμε από την τεχνογνωσία και πραγματογνωμοσύνη των ΗΠΑ. Για παράδειγμα το EPA τώρα θέτει προδιαγραφές σαφείς για την καθαρή ατμόσφαιρα όσον αφορά την διαρριγμάτωση και τις τεχνολογικές δυνατότητες και απαιτούν, ζητούν 95% των εκπομπών ρήπων θα πρέπει να συλλαμβάνονται και να αποθηκεύονται. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον όλα αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να τα εμπεριέχουμε και να τα συμπεριλάβουμε σε αυτά που θεωρούμε ότι είναι αποδεκτά και πρέπει να προσφέρονται στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Σιμάνσκι τελευταίος ε, σκιώδης ηγητής. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Θα προσπαθήσω βέβαια. Πρώτα, ευχαριστίες μου προς την κυρία Συγχύτρια για τον διαφανή τρόπο και ανοιχτό τρόπο διατύπωσης έκθεσης. Τώρα, σε σχέση με τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Μπουτικόφερ, συμφωνώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την αμερικανική πραγματογνωμοσύνη και πείρα. Και τουλάχιστον τμήμα αυτής είναι το ότι υπάρχει μόνο μία μελέτη. Η μελέτη Φόρτς που δείχνει, καταδεικνύει ότι το ίχνος των εκπομπών ρήπων του σχιστολιθικού αερίου είναι υψηλότερο από το ίχνος άνθρακα στην ατμόσφαιρα και αυτό σε σχέση με τις χαμηλές υποδομές τεχνολογικών ρωσικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τους Ρώσους για το διοξίδιο του άνθρακα και άλλες εκπομπές ρήπων. Η Αμερικανική λοιπόν πείρα δείχνει ότι υπάρχει καθαρή λύση που προσφέρεται για τις χώρες που βρίσκονται υπό την εξουσία του άνθρακα σήμερα, εξαρτώνται από τον άνθρακα. Και η δυνατότητα διαρριγμάτωσης ε, χωρίς χημικές ουσίες. Το να προτείνουμε κάτι τέτοιο είναι το να προτείνουμε να υπάρχουν ανεμόμυλοι χωρίς άνεμο. Είναι ίσως ε, κάτι που θα μπορούσαμε να υποσχεθούμε αλλά δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Για τις παρατηρήσεις για τη Βουλγαρία τώρα. Στη Βουλγαρία δεν υπάρχει κανένας ε, καμία πορεία, κανένας δρόμος, κανένας τρόπος που θα ισοπεδώναμε κανέναν. Ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε η Βουλγαρία να απόσχει από αυτές τις επενδύσεις είναι τελείως διαφορετικός. Δεν είναι το κοινωνικό πρόβλημα με το railroading, δηλαδή την ισοπαίδωση και αγνόηση των πολιτών. Αλλά επανερχόμενος στο σχιστολιθικό αέριο και σχιστολιθικό πετρέλαιο είναι θέμα δικού μας δυναμικού και γι' αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε αυτά τα θέματα διότι δεν ε, είμαστε πλούσιοι με τέτοιου είδους πόρους και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε γρήγορση για τη διάθεσή τους στην αγορά. Σίγουρα αυτό θα σημαίνει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Σίγουρα μεγαλύτερος ανταγωνισμός θα σημαίνει καλύτερες τιμές, καλύτερες προϋποθέσεις και προσφορές για τους πολίτες και για τις βιομηχανίες. Τώρα, οι συμπτώσεις ε, και η, ε, και σύγκληση για τους πολίτες και την υλοποίηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την παρουσία αυτών των προϊόντων στην αγορά. Πολύ καλή συγκυρία ενισχύει και ενδυναμώνει τη συγκυρία και τη συνέργεια που θα βοηθούσε την μεγαλύτερο ε, ανταγωνισμό στις αγορές μας. Πολλοί ανησυχούν για τον όγκο των πόρων μας, του δυναμικού μας. Δεν είναι δική μας δουλειά εμείς οι πολιτικοί να αποφασίσουμε το σχήμα ή μορφή οποιασδήποτε ε, εξέλιξη στην αγορά ενέργειας. Είναι θέμα γεωλογίας και επενδυτών να αποφασίσουν τι είναι οικονομικά εφικτό, τι είναι εμπορικά κερδοφόρο και σημαντικό. Εμείς ως πολιτικοί ο ρόλος μας δεν είναι να, υπονομεύσουμε αυτές τις δραστηριότητες και να δούμε τις δυνατότητες ε, όχι μόνο για την εξέλιξη αυτή αλλά και για μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άλλες πέντε τοποθετήσεις υπάρχουν. Παρακαλώ τους συναδέλφους να σταθούν στα δύο λεπτά. Γιατί έχουμε ακόμη ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Και έχουμε και, με... και σύντομες πληροφορίες να σας δώσουμε για το τι διεμήθη χθες τους συντονιστές. Παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Ο κύριος Μαρτσινκίεβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα και πάλι ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που θα είναι σημαντική για τις αναδυόμενες αγορές για το μέλλον. Θα έπρεπε για όλους αυτούς τους λόγους να αντιμετωπίσουμε όλες τις πηγές ενέργειας ισότιμα και ισοδίκαια. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε, πιστεύω, ένα πρόγραμμα ένα πρόγραμμα υποστήριξης ε, της έρευνας ώστε να μπορέσουμε να αναλύσουμε και να δούμε ποια είναι τα αποθέματα σχιστολιθικού αερίου στην Ευρώπη και δεδομένης της κοινή ενεργειακής αγοράς για την ανάπτυξη της ενεργειακής αυτής αγοράς έχει τη σπουδαιότητά του αυτό το θέμα. Βλέπουμε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ από την άλλη πλευρά και ίσως θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνολογίες χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον λοιπόν και αυτό θα ήταν τεράστια σημασία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την άλλη πλευρά και μια σύντομη άλλη παρατήρηση. Θα ήθελα να προσθέσω το ανέφερε αυτό ο κύριος ε, Ρούμπικ και ο κύριος Ρούμπικ Μπιουτικόφερ. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την παραγωγή ενέργειας ε, ηλεκτρικού ρεύματος από την εκμετάλλευση άνθρακα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε επαρκείς μονάδες αερίου. Αυτό θα πρέπει να επιδιώξουμε. Το ίδιο ισχύει για όλους εκείνους που κάνουν λόγο για τις πράσινες περιβαλλοντικές πηγές ενέργειας. Η μόνη εναλλακτική δυνατότητα για να μην σταματήσει να λειτουργεί το σύστημα είναι το φυσικό αέριο. και πρέπει το φυσικό αέριο να λάβουμε υπόψη για την παραγωγή αυτής της ενέργειας που χρειαζόμαστε. Ε, Madame please. Κυρία Κολάσκα Μποβίσκα παρακαλώ. Thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ζαβέλα για την έκθεσή της. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή έκθεση. Δεύτερον, πιστεύω ότι στην δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή θα προετοιμάσουμε και θα καταθέσουμε τροπολογίες. Θα έπρεπε να καλύπτουν το θέμα της έκθεσης που είναι η αγορά ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Επειδή οι περιβαλλοντικές πτυχές βρίσκονται συζήτηση και σήμερα και αύριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβού της Ευρωβουλής. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στο κύριο θέμα της έκθεσης ε, και όχι σε άλλα. Τώρα, στρέφομαι σε περισσότερο εξειδικευμένα θέματα. Όπως και προανέφεραν κάποιοι συνάδελφοί μας, ε, το 2030 δεν είναι ρεαλιστικό στόχος ως ημερομηνία για το συστολιθικό αέριο ως ε, πηγή ενέργεια δεν είναι όμως ε, εξωρεαλιστική, εξωπραγματική για την Πολωνία που ξεκινά την εξόριξη το 2014 νομίζω. Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση μέχρι το 2016 ή 2017, αλλά μέχρι τότε θα είναι ευδιάκριτη πρέπει να πω. Δεν είναι λοιπόν εξωπραγματικός αυτός ο στόχος για μας, για την Πολωνία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα είναι οι κοινωνικές αντιδράσεις. Ο κύριος Μπιουτικόφερ ανέφερε τις αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιες χώρες. Κύριε Μπιουτικόφερ, ταξίδευα εγώ στην περιοχή Λουμπέσκα, όπου υπάρχει μεγάλη πυκνότητα δραστηριοτήτων συστολιθικού αερίου. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι πολλές διαμαρτυρίες κατά του φυσικού αερίου και κατά της αιωλικής ενέργειας είναι πολύ εντονότερες από ότι οι διαμαρτυρίες κατά του συστολιθικού αερίου. Αυτό λοιπόν που μπορώ εγώ να σας πω και να τεκμηριώσω είναι ότι οι πολίτες, οι πολίτες απλά φοβούνται. Δεν γνωρίζουν πολλά για νέες πηγές ενέργειας και το συστολιθικό αέριο είναι μόνο μία από αυτές τις νέες πηγές ενέργειας. Η πράσινη ενέργεια είναι μία νέα πηγή ενέργειας για αυτούς. Είναι κατανοητό να υπάρχουν φοβίες έναντι αυτών των πηγών ενέργειας όσο σε σχέση με το συστολιθικό αέριο για παράδειγμα αναγκαίο είναι αυτές οι πτυχές σε σχέση με αυτά τα θέματα να διασφαλίσουμε ότι θα είναι φιλο, ε, φιλικές προς το χρήση και να δούμε τι θα πρέπει να γίνει. Είναι θέμα κατανόησης. Είναι θέμα του να δώσουμε διασφαλίσεις στους πολίτες μας ότι κάποιες αρχές μεριμνούν για την ασφάλειά τους μεριμνούν για την ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού στο νερό, σε νερό, σε θέματα περιβαλλοντικά που διασφαλίζουν. Αυτό είναι αναγκαίο σε σχέση με τα θέματα αυτής της έκθεσης. Είναι πολύ σπουδαία αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωσέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω μερικές παρατηρήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά στο αέριο που κατά την παράγραφο 9 της έκθεσης θα έχει λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ότι ο άνθρακας ή το πετρέλαιο. Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι άμα δούμε συνολικά το αέριο, όχι μόνο δηλαδή την εξαγωγή του και την κατανάλωσή του αλλά και τη μεταφορά του και την επεξεργασία του έχουμε πολύ λες περισσότερες διαφυγές από ότι με το πετρέλαιο και τον άνθρακα και το οικολογικό του χνάρι για την παραγωγή φαινομένου του θερμοκηπίου ε, είναι συγκρίσιμο αν όχι μεγαλύτερο με τις άλλες ορυκτές πηγές ενέργειας. Το στο λιθικό αέριο λοιπόν είναι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο και από το φυσικό αέριο. Επίσης, ε, μία ε, επιστημονική αμερικάνικη μελέτη αποδεικνύει ότι στα κεντρικά κράτη, στις κεντρικές πολιτείες ε, των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Τακότα μέχρι το Τέξας αυτή η υδραυλική γεώτρηση οδηγεί σε μία αύξηση των σεισμικών επεισοδίων δεν είναι μόνο το νερό το οποίο μολύνεται, αλλά και σεισμογραφικά ε, ε, έχουμε μεγαλύτερα σεισμογραφικά φαινόμενα όταν χρησιμοποιούμε την υδραυλική γεώτρηση για την εξαγωγή του σχιστολιθικού αερίου πρόκειται για μεθάνιο, δεν είναι διοξίδιο του άνθρακος. Οπότε η ραδιενεργός πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη και ρηπαντική. Τώρα σε επίπεδο βιομηχανικό και οικονομικό, όπως ξέρετε για, τον, για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, ε, η εκμετάλλευση στο χρονικά ε, δεν έχει διάρκεια. Μέσα σε δύο χρόνια έχετε βγάλει το 80% της γεώτρησης και πρέπει κάθε φορά να ε, προχωρείτε σε γεωτρήσεις βαθύτερες, βαθύτερες, βαθύτερες. Και δεν είναι σίγουρο ότι μακροπρόθεσμα, διότι πέντε χρόνια υπάρχει ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είναι εγγυμένο λοιπόν μακροπρόθεσμα ότι η παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου θα κρατήσει στο χρόνο. Η κυρία Ήμπνερ. χωρίς μικρόφωνο. Ε, ευχαριστώ την κυρία Τζαβέλα για την επαγγελματικότατη προετοιμασία του δύσκολου αυτού θέματος. Υπήρξε πολύ λογική στην προσέγγιση της. Από τη μία εξέτασε τη βιομηχανική πτυχή και από την άλλη τόνισε και το θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι γεγονός ότι πρέπει να τα δούμε όλα από κοντά και τώρα που σε μερικές χώρες έχει αρχίσει η εξόριξη και εν ώψη νέων εξορίξεων. Επίσης, υπάρχει διαδεδομένος φόβος, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά για να ησυχάσουμε τον κόσμο μπροστά σε αυτούς τους φόβους. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης των πόρων που σημειώνεται στην Ήπειρό και θα θέλαμε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τις ενεργειακές ανάγκες, τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Χρειάζεται ίσως περισσότερη έρευνα. Θέλουμε να μειώσουμε ή να καταργήσουμε, να σταματήσουμε τους πυρηνικούς σταθμούς ή όχι. Πολλοί δεν ικανοποιούνται από αυτή τη λύση της πυρηνικής ενέργειας γιατί λένε ότι τα πυρηνικά απόβλητα είναι ορολογιακή βόμβα. Ίσως πρέπει όντως να την παρατήσουμε. Όσο για τις προτάσεις που συζητάμε σήμερα, πρέπει όλες οι χώρες να μπορέσουν να απλοποιήσουν και να εκλογικεύσουν τον τρόπο παραγωγής ενέργειας που διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Για την οικονομία με λιγότερο άνθρακα μέχρι το 2050, αυτό εννοεί ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλο και λιγότερο, να χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερο τον υπάρχοντα άνθρακα, άρα πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να δούμε αν γίνεται να αντικαταστήσουμε τον άνθρακα με κάτι άλλο από τις χώρες μας. Αλλιώς θα χρειάζεται ακόμη να εισάγουμε πετρέλαιο και άλλες ενεργειακές πηγές. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία εισηγήτρια για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα που μας παρουσίασε. Ευχαριστούμε κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και εγώ θέλω να κάνω μια προειδοποίηση, να ζητήσω φρόνηση δηλαδή. Διότι Είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε πηγάδι αργά ή γρήγορα θα σταματήσει να βγάζει νερό. Και το ίδιο ισχύει και για τους πιστόλιθο. Είναι πεπερασμένη και αυτή η πηγή και υπάρχει και ο φόβος των χημικών και της ε, διάχυσής τους στο περιβάλλον. Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα. Εγώ δεν θέλω να αντιταχθώ ως θέμα αρχής στο θέμα της εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού αερίου. Θέλω να γίνει απλώς μια σύγκριση της μεθόδου αυτής που υπάρχει με άλλες μεθόδους παραγωγής αερίου. Παραδείγματο χάρη τα αγροτικά απόβλητα ή τα δασοκομικά απόβλητα. και τη μόλυνση που υπάρχει γύρω από όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και από βιομάζα, βλέπουμε ότι όλες οι πηγές παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να τις συγκρίνουμε. Αναρωτιέμαι αν πρέπει ή όχι να εκμεταλλευτούμε παραπάνω το σχιστολιθικό αέριο, γιατί υπάρχει και το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών δεν νομίζω ότι πρέπει να βιαστούμε γιατί είναι και αυτή η καταστροφική μέθοδος για το περιβάλλον και την οικολογία. Δεν θέλουμε να χειροτερέψουμε τα πράγματα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν την εκμετάλλευση αυτή γιατί έχουν πολύ λιγότερη πυκνότητα πληθυσμού. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά και είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Κομισιόν τώρα, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αλλά σύντομα γιατί καθυστερούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι όντως συντοπάτατος. Γνωρίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε και προς το τελευταίο θέμα. Εμείς από την Κομισιόν ε, εγκρίνουμε την έκθεση αυτή και ενδιαφερόμαστε για τη συζήτηση του Κοινοβουλίου για το σχιστολιστικό αέριο. Είναι ένα θέμα που και η Κομισιόν, που ενδιαφέρει και την Κομισιόν όταν λέω χαιρόμαστε για την έκθεση αυτή εννοώ ιδιαίτερα διότι τονίζει τη σημασία που έχει η συμπλήρωση της ενιαίας της εσωτερικής αγοράς. Κατ' εμάς είναι πράγματι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλουμε και η νέα αυτή πηγή αερίου να συμπεριλαμβάνεται στις πηγές που διαθέτουμε. Επίσης με ικανοποίηση ακούσαμε ότι η συζήτηση αυτή για το σχιστολιθικό αέριο είναι μέσα στα πλαίσια της συζήτησής μας για την οικονομία χωρίς άνθρακα μέχρι το 2050. Όσο για το, κατα... πόσο σχιστολιθικό αέριο μπορούμε να παραγάγουμε, κάνουμε μία μελέτη αυτή τη στιγμή και θα... τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σε λίγο ελπίζουμε πριν τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Ακούστηκαν πολλά για διάλογο με τους πολίτες και για τις ανησυχίες των πολιτών. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε τη χρήση κονδυλίων για να το μελετήσουμε και αυτό. Τέλος, το θέμα των αερίων με εφέ θερμοκηπίου. Σε σύγκριση με άλλα καύσιμα ως προς το σχιστολιθικό αέριο. Και εδώ γίνεται μια μελέτη η οποία και αυτή θα δημοσιευτεί σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Είχαμε ξεχάσει το συνάδελφό μας Έλμερ για ένα λεπτό. Κοιτάξτε, δεν μιλήσαμε καθόλου για την ανταγωνιστικότητα των εφορών ενεργειακών πηγών. Υπάρχει Κίνα, υπάρχει Ινδία που έχουν εκατοντάδες σταθμούς, ε, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα και αποτελούν μια ανταγωνιστική για μας πηγή ηλεκτρικής ενεργείας, φτηνότερη μάλιστα. Εμείς εξαρτώμαστε τώρα πια όλο και περισσότερο από τις ανανεώσιμες. Έχουμε δυνατότητες μείωσης και των πηγών και των τιμών χρησιμοποιώντας τις πηγές που υπάρχουν τοπικά αντί να σκεφτόμαστε όνειρα όπως την αιωλική ενέργεια. Γιατί εδώ είναι η ομάδα πίεσης των πρασίνων που αντιδράει συνήθως ιστερικά κατά η, της πυρηνικής ενέργειας παραδείγματος χάρη. Ε, ας περιμένουμε αν είναι έτσι μέχρι να μην μπορούμε να παράγουμε καθόλου ηλεκτρισμό. Πρέπει να καθησυχάσουμε και το κοινό. Είναι και αυτό καθήκον μας, διότι το κοινό αυτό ε, γίνεται αντικείμενο προπαγάνδας από τους πράσινους. Γίνεται θύμα προπαγάνδας από τους πράσινους. Αυτά που λένε για τους σεισμούς, για τις... Ε, εξορίξεις, για τα ανθρακοριχεία. Δεν είναι όλα αυτά αληθινά. Πρέπει να τα εξεχωρίσουμε τα σωστά από τα λάθη. Ευχαριστώ. Κυρία Τζαβέλα, 30 δευτερόλεπτα σας παρακαλώ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά μακροσκελής έκθεση. 30 δευτερόλεπτα σας παρακαλώ στα συμπεράσματα. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Θα ήθελα να πω ότι σε όσα ελέγχθησαν και υπάρχουν ενδιασμοί, υπάρχουν τεχνικές απαντήσεις το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, θέλω να υπενθυμίσω, οι οποίες είναι στη διάθεσή σας, μου δίνετε 30 δευτερόλεπτα, εν Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις χώρες που έχουν σε gas να προχωρήσουν, γιατί αν δεν προχωρήσουν δεν θα δούμε και τι επιπτώσεις έχει. Ξέρουμε καλά ότι πάμε εκ του ασφαλούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δεχθούμε τους ενδιασμούς που υπάρχουν. Και το τρίτο είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να τολμήσει και να προχωρήσουμε να αξιοποιήσουμε τις δικές μας πηγές. Είμαστε αρκετά μεγάλοι ως Ευρώπη και αρκετά όριμοι για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και την υγεία του πληθυσμού μας. Μόνο αν προχωρήσουμε θα ξέρουμε πώς θα προστατεύσουμε και την υγεία του πληθυσμού μας. Κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει κακό στις τοπικές κοινωνίες. Όλη η πληροφόρηση που έχω είναι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 8 Μαΐου στις 12. Τελειώνουμε με αυτό το σημείο. Επόμενο σημείο. Δίνω το λόγο στον Καστόν ε, Φράνκο για το LIFE, το πρόγραμμα για το περιβάλλον και για το κλίμα. Oui, merci, euh, la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα κοιτάξω να προχωρήσω γρήγορα, αλλά νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα LIFE ε, χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Θα σας παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου. Εγώ πρότεινα 19 τροπολογίες ε, γύρω από αυτό το θέμα που είναι επικεντρωμένο σε θέματα περιβάλλοντος. Αποτελεί πρόκληση για την Επιτροπή Βιομηχανίας, ε, η, Περιφερειακή, η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και ο προπολογισμό επίσης πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Θέλει να δημιουργήσει ένα ειδικό μέσο για, την, ε, για το περιβάλλον η Κομισιόν για το 2014-2020. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ικανοποίησε μέχρι τώρα τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει όμως να βελτιώσουμε το feedback. Ε, η χρηματοδότηση του Natura 2000 από το πρόγραμμα LIFE και αποτέλεσε ε, πηγή πειραματικής καινοτομίας ε, το LIFE. Συνέβαλε στη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας για το περιβάλλον στην Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει η Κομισιόν συμβαδίζει περισσότερο με τις προκλήσεις για το περιβάλλον της ε, εποχής μας και προβλέπει και μία δράση για το κλίμα. Πρώτο σημείο της νομοδότησής μου είναι η αντίληψη του ολοκληρωμένου σχεδίου. Πρόκειται για τη βασική πρόκληση του νέου προγράμματος χρηματοδότηση περιβαλλοντικών και κλιματικών προγραμμάτων με συνολική περιβαλλοντική προσέγγιση βασιζόμενη στη συνέργεια των κοινωτικών κονδυλίων, των εθνικών μέσων και των προσθετικών μέσων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η ιδέα της ε, ταμιοποίησης είναι ε, σωστή. Μπορούμε να φανταστούμε τη χρηματοδότηση των τοπικών σχεδίων για το κλίμα. Πώς θα λειτουργήσει όμως κάτι τέτοιο στην πράξη. Οι διαδικασίες, τα χρονοδιαγράμματα, οι συνθήκες των διαφόρων ταμείων δεν είναι ταυτόσιμα και η συμπληρωματικότητα δεν λειτουργεί σε όλο τον, τους κανονισμούς των ταμείων. Τι εγγύσεις η Κομισιόν λοιπόν σκοπεύει να δώσει για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των συνολικών σχεδίων. Για, τις, για την γεωγραφική ισορροπία των ολοκληρωμένων σχεδίων θα έπρεπε να διευκρινιστεί η πρόσταση της Κομισιόν στο Κοινοβούλιο. Πρέπει το ΛΑΙΦ να καταστεί η πραγματική βιομηχανία φυσικού αερίου, μιλούσαμε προηγουμένως, ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος, η προστασία και ε, αποκατάσταση της βιοπικιλότητας θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό στόχο. Θα πρέπει να ενσωματωθούν όμως και δράσεις για την καταπολέμηση του θορύβου ή για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να ε, στοχεύει να ε, παρέμβει και στον τομέα των υδάτων. Εγώ θα ήθελα όμως να δοθεί με περισσότερη ακρίβεια το τι θα γίνει με το θαλάσσιο περιβάλλον. Τώρα, για, την, ε, για το κόστος της ε, καινοτομίας. Το LIFE θα πρέπει να χρηματοδοτήσει οικοκαινοτόμες δράσεις και αυτό στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ορίζοντας 2020. Θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έτσι πειραματικές προσεγγίσεις για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών και νέων ε, μεθόδων για το κλίμα και το περιβάλλον. Αυτό θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την αριστεία τους και κυρίως τις ΜΜΕ. Γεωγραφική κάλυψη του LIFE. Χαίρομαι που στο άρθρο 5 του κανονισμού μπορούμε να χρηματοδοτούμε σχέδια στις γειτονικές χώρες στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, διότι με αυτές τις χώρες συμμεριζόμαστε κοινέ περιβαλλοντικές προκλήσεις. Λυπούμε όμως που οι πόντιες περιφέρειες ε, δεν συμπεριλαμβάνονται. Θα, ε, ε, θα ήθελα το BEST, η προστασία δηλαδή της βιοποικιλότητας, να εφαρμοστεί και στις υπερπόντιες περιφέρειες της Ένωσης. Και θα έπρεπε να έχουμε και ένα μάξιμουμ ε, στις ε, χρηματοδοτήσεις για να μην έχουμε ε, σπατάλες. Για την επιλεξιμότητα του κόστους θα έπρεπε να έχουμε ένα γενικό προβληματισμό για την επιστροφή του ΦΠΑ συνολικά για τα προγράμματα διαποντέ από τον δημοσιονομικό κανονισμό και όχι μόνο από το πρόγραμμα LIFE. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας σχετικά. Σχετικά με την επιλεξιμότητα και το κόστος του μόνιμου προσωπικού πρέπει να... Εγώ το σκέφτομαι διαφορετικά από την Κομισιόν. Ε, θα έπρεπε αυτές οι δαπάνες να συνεχίσουν να επιστρέφονται για να μην επιβαρύνουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία είναι ιδιαίτερα εμπλεγμένη στο νέο πρόγραμμα LIFE. Ευχαριστώ συνάδελφε Φράνκο και για την κατανόησή του για το χρόνο. Αυτό το πρόγραμμα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Άρα θα το ξανασυζητήσουμε όταν θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Η συνάδελφος Βαμπρέντ που είναι σκιώδης εισηγήτρια. Κάθριν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και μετά θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ το ίδιο σύντομη και τηλεγραφική για να μπορέσουν να μιλήσουν και άλλοι στα επόμενα πέντε λεπτά που μας έχουν μείνει. Το πρόβλημα του προγράμματος Life είναι ο προπολογισμός του. Δεν είναι εύκολο να ζητήσουμε περισσότερα κονδύλια βέβαια, αλλά εγώ είμαι μεν υπέρ τέτοιων αυξήσεων, αλλά πρέπει να το δούμε και γενικότερα. Υπάρχει ο προϋπολογισμός της γεωργίας, της υπέθ, του υπαίθριου χώρου κτλ. Πρέπει να το δούμε λοιπόν γενικότερα και να σκεφτούμε τις δημοσιονομικές προοπτικές. Δεύτερον, η ομάδα μας είναι υπέρ των ολοκληρωμένων ταμείων. Στον προϋπολογισμό παραμένουν ακόμη πολλά προβλήματα προσωπικού, ΦΠΑ. Πρέπει άρα πρώτα να ξεκαθαριστούν τα πράγματα και να διαχωρίσουμε τις μη κυβερνητικέ αργανώσεις από τις δημόσιες αρχές, διότι δεν θα πληρώσουμε τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών με τα ελάχιστα χρήματα που διαθέτουμε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό υπαλλήλου των χωρών με δημοσίους υπαλλήλου ή μήκη όμικρον. Συμφωνώ με τον εισηγητή τέλος ότι η Κομισιόν πρέπει να αναφέρει και τις διάφορες οι ε, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Ένωση οικοκαινοτόμες γιατί θέλουμε πολύ καινοτομία Ιδίω ως προς το περιβάλλον και το live εδώ θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο υποστηρικτικό. Ευχαριστούμε την κυρία Βαν Πρέντ Φιουνάουλ. Ευχαριστώ. Και εγώ τον εισηγητή θα παραμείνω και εγώ σύντομη. Πρώτον συμφωνώ ότι το live υπήρξε επιτυχές και πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσε να τύχει καλύτερης δημοσιότητας, περισσότερης. Για τον προϋπολογισμό νομίζω ότι μέσα στους περιορισμούς που μας θέτουν οι δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός του live θα προστατευτεί, θα παραμείνει και δεν θα χαθεί μεταξύ των υπολείπων πυρικοπών. Δεύτερον, δεν έχω πιστεί ούτε η ίδια για τα ολοκληρωμένα λεγόμενα προγράμματα. Θέλω να ακούσω και τους άλλους, αλλά έχω μερικές ανησυχίες προς το κατά πόσον προσθέτουν τίποτα. Μπορεί απλώς να υπάρχει επικάλυψη, άχρηστη επικάλυψη. Συμμερίζομαι την ανησυχία του εισηγητή ότι μπορεί αυτά τα λεγόμενα ολοκληρωμένα προγράμματα να αποτελέσουν κάποιο κατακαιρματισμό των αρχικών στόχων του LIFE. Τέλος, συμφωνώ ότι ότι αυτά που λέμε στη χώρα μου ως τι πρέπει να συσχετιστούν και αυτά. Γιατί μερικές χώρες έχουν πολύ μεγάλη βιοπικιλότητα και δεν έχει νόημα στην Καραϊβική μερικά νησιά να, έχουν, να την χάνουν όσοι τι και άλλες χώρες όχι. Και εδώ στηρίζω την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κωσέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής και η Κομισιόν μας ανέφεραν σωστά πράγματα, ιδιαίτερα την δημιουργία του υποπρογράμματος για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Επίσης εξετίμησα ιδιαίτερο στο σκεπτικό 14 που παραλληλίζει την προστασία των δασών με την ικανότητα απορρόφησης του διοξιδίου. Είναι λοιπόν μια οικολογική συστημική προσέγγιση. Ο συνάδελφος Φράγκο έκανε μια έκθεση με πολύ σωστά σημεία και θα υπερψηφίσουμε και πολλές από τις τροπολογίες του ιδιαίτερα για τη συμπερίληψη των υπερποντίων διαμερισμάτων που έχουν ιδιαίτερη χλωρίδα και πανίδα. Στις νησιωτικές πολλές φορές αυτές περιοχές. Και στο 10 και στο 11 λέει πολύ σωστά πράγματα. Προσθέτει την έννοια του οικολογικού διαδρόμου Συμφωνώ και εγώ κύριε Σιγητά ότι οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα οι μικρότερες μήκη ο δεν έχουν αρκετή χρηματοδότηση 0,3% είναι κάτι πολύ χαμηλό αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει κρίση θα θέλαμε βέβαια παραπάνω τέλος πάντων λυπάμαι γιατί δεν υπάρχει καθόλου το θέμα των όλο και λιγότερων πρώτων υλών. Το είπαμε λίγο γενικά προηγουμένως για το πετυρέλαιο, αλλά υπάρχουν και άλλες μη ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και η μελλοντική τους σπάνιθ θα γίνει, θα όλο και περισσότερο προβληματική. Πρέπει να το προσθέσουμε αυτό υπάρχει και η έκφραση οικονομία με χαμηλή ανθρακοεντατικότητα. Εδώ υποψιάζομαι ότι η έκφραση αυτή υπονοεί πάντοτε την πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων. Γενικά είμαι αρκετά υπέρ της έκθεσής σας κύριε συγητά μου. Αν και στο 16 επαναλαμβάνω του σκεπτικού, τίθεμαι κατά της προώθησης της αποθηκεύσεως του διοξιδίου. Δεν υπάρχουν άλλοι σκιώτες. Ο συνάδελφος Έλμερ. Παρακαλώ να είναι σύντομος. Δεν έχω τίποτα προσωπικό εναντίον του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και επίσης συγχαίρω και εγώ την εισηγήτρια και για την βιοπικιλότητα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να υποστηρίξουμε τις προτάσεις. Όμως απογοητεύουμε τόσο μεγάλη, ε, μεγάλο μέρος της έκθεσης και του προϋπολογισμού βασίζεται στις, ε, του σειρμού αιμονές μας για το πρασίνισμα. Κάνω λόγο για τις κλιματικές αλλαγές. Γνωρίζουν οι συνάδελφοι το εύρος ε, των αλλαγών όπου πολλοί επιστήμονες κρούν κόδωνα κινδύνου εφιστώ την προσοχή στον James Lovelock, αυτόν τον γκουρού, τον παππού της περιβαλλοντικής κίνησης, τον ε, ε, εφευρέτη της έννοιας της ε, γέας που έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι οι κλιματικές αλλαγές θα σκοτώσουν, θα δολοφονήσουν την ανθρωπότητα με κάποιες εξαιρέσεις στο Βόρειο και Νότιο Πόλο. Γνωρίζουν συνάδελφοι ότι δημοσίευσε ένα βιβλίο πρόσφατα που λέει ότι κάναμε λάθος. Υπερτονίσαμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο κακό. Πριν από 20 χρόνια νομίζαμε ότι γνωρίζαμε τι θα έκανε το κλίμα. Τώρα αναγνωρίζουμε ότι κάναμε σφάλμα. Ε, λοιπόν, γίνονται σφάλματα και σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο για τους ίδιους λόγους. Ευχαριστώ. Grazie. Ε, Ευχαριστώ τους ε, μεταφραστές για την κατανόησή τους. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και μετά ο συνάδελφος ε, Φράνκο για τα συμπεράσματα. Δύο εκπρόσωποι της Κομισιόν είμαστε εδώ. Εγώ εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η συνάδελφος Μετεκουίν ασχολείται με το κλίμα. Ευχαριστώ τον κύριο Φράνκο για το σχέδιο έκθεσης, αλλά και τους βουλευτές που πήραν το λόγο και θα ήθελα ε, στα πλαίσια των συζητήσεων που έγιναν να υπογραμμίσω μερικά σημεία και να αντιδράσω πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο την κυρία Κουίν Συγγνώμη, έχετε μόνο ένα λεπτό Είμαστε εκτός χρόνου, ωραία, πολύ σύντομα ο κύριος Φράγκο υπογράμμισε ορισμένα σημεία, τα ολοκληρωμένα σχέδια ήταν το πρώτο σημείο, όπως είπαμε το πρόγραμμα LIFE δεν έχει μεγάλα, ε, με μεγάλο φάκελο, χρηματοπτικό φάκελο. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το LIFE ως μοχλό των άλλων ε, σχεδίων, των άλλων προγραμμάτων ε, και να βοηθήσουμε την Κομισιόν ε, να ε, εφαρμόσει καλύτερα την νομοθεσία για το περιβάλλον. Ε, υπογραμμίστηκαν μερικά μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών και όπως και το Ταμείο Συνοχής. για τα κοινά στρατηγικά προγράμματα που συντονίζουν την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών και κομισιών γίνεται αναφορά στο LIFE αλλά και σε άλλα προγράμματα στην ΚΑΠ και εκεί θα, κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις των δημοσιονομικών προπτικών το κοινοβούλιο να ε, επιμείνει ούτως ώστε να αναφέρεται το live. Για τα θέματα ε, εφαρμοστικού πεδίου του ολοκληρωμένου σχεδίου λέγεται ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θόρυβο και με το αστικό περιβάλλον και το νερό. Θυμίζω στο Κοινοβούλιο ότι ο δημοσιονομικός φάκελος είναι πολύ μικρός ε, και μόνο αν αυξηθεί ο προπολογισμό μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η δημοαρχή του προπολογισμού θα πρέπει να αποφασίσει το Κοινοβούλιο. Επίση, ανοίξει από την αρχή, μπορεί να κάνει κάτι. Για τι υπερπόντιε περιοχέ δεν αναφέρονται ειδικά στο live. Η οι υπερπόντιες περιοχές ε, λογικά θα πρέπει να καλύπτονται από το LIFE. Υπάρχει μία απόφαση σχετικά και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται ειδική αναφορά στις υπερπόντιες περιοχές. Στον κανονισμό για την επιλεξιμότητα του κόστους ε, καλό είναι να γίνεται αναφορά στον δημοσιονομικό κανονισμό που διαπραγματευόμαστε σήμερα ε, για την τριετία αναθεώρηση και σε αυτόν τον κανονισμό, δεν ξέρω ίσως η συνάδελφο, συγγνώμη, συγγνώμη, πραγματικά. Ε, κυρία Κουίνε, ζητώ πραγματικά συγγνώμη, αλλά σας παρακαλώ να στείλετε στον εισηγητή και στους άλλους και όδης τις παρατηρήσεις σας γραπτός, διότι θα ήθελα αυτά τα τρία λεπτά που μας μένουν να τα πείσω στον εισηγητή. Σας παρακαλώ να στείλετε γραπτός τις παρατηρήσεις. Λυπούμε, λυπούμε για την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Αλλά έχουμε πρόβλημα ωραρίου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους εκπροσώπους της Κομισιόν για τη θετική του συνεισφορά. Τα προβλήματα προϋπολογισμού τα σημεριζόμαστε. Θέλω να διασφαλίσω τη συνάδελφο για τα ολοκληρωμένα σχέδια. Δεν αντικαθιστούν τα υπάρχοντα σχέδια, αλλά λειτουργούν προσθετικά. Ε, δίνουμε εμείς εδώ έναν άλλο τρόπο εργασίας ε, που θα πρέπει να αρχίσει να ροντάρει. Ελπίζουμε αυτό το φαινόμενο μοχλός να λειτουργήσει, του live δηλαδή να λειτουργήσει στα άλλα προγράμματα. Και κυρία Πρόεδρε, μην μπείτε στην Γαλλία ότι συμμερίζομαι τις πράσινες ψυχώσεις του Ιβ Κοσέ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών 26 Απριλίου στις 12. Ολοκληρώνοντας, αναφέρω για τη συνεδρίαση των συντονιστών και λέω ότι τρεις αντιπροσωπείες Οι τρεις αντιπροσωπείες που θα πάνε στις διάφορες επισκέψεις θα οριστούν από τους συντονιστές που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις ομάδες και το συσχετισμέ τους. Επίσης, ε, εκθέσεις Energy Star στους μη εγγεγραμμένους, η συμφωνία με την Αλγερία με απλουστευμένη διαδικασία από το Προεδρείο για τη γνωμοδότησή μας για την ΚΟΠΑ 18, το πήραν οι σοσιαλιστές και η γνωμοδότηση για την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπή της Ρέτζη για τα Ταμεία Συνοχής και τις Ενεργειακές Πολιτικές και το ρόλο τους. Δόθηκε επίσης στους σοσιαλιστές που είχε τους πόντους. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Συγγνώμη κυρία Κουίν, ξέρετε ότι το ένα λεπτό είναι ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ όλους.